nie możemy sobie pozwolić na dłuższe opóźnienie niż pięciominutowe. Καλημέρα σας. Ε, καθυστερήσαμε κάτι παραπάνω. Ας μην χάσουμε άλλο χρόνο. Και θα ήθελα κυρίες και κύριοι να σας ενημερώσω ότι για τα πρώτα 15 λεπτά το Europal TV θα μαγνητοσκοπεί την συνεδρίασή μας για να αξιοποιήσει, χωρίς ήχο, για να αξιοποιήσει το υλικό για το έργο των Ευρωβουλευτών. Θα είναι λοιπόν μόνο μαγνητοσκόπηση, μόνο βίντεο. Αυτό για να είστε ενήμεροι. Σφαλώς θα έρθουν και άλλοι συνάδελφοι σε λίγο. Έχετε την ημερήσια διάταξη. Αντιρρήσεις δεν φαντάζομαι να υπάρχουν. Έχουμε 19 γλώσσες εκτός από τσεχική, μαλτεζική, σλοβακική, σλοβενική και γκέλικη, ιρλανδική. Θα μιλήσουμε για το μέλλον των τροφίμων και της γεωργίας, αυτό είναι το σημερινό μας θέμα, με εισηγητή τον κύριο Ντόρφμαν. Σήμερα θα γίνει ουσιαστική συζήτηση, κύρια συζήτηση του θέματος. Το έχουμε συζητήσει βέβαια πολλές φορές, γιατί δεν υπάρχει συνεδρίαση της Επιτροπής μας που να μην συζητείται το μέλλον ε, της ε, γεωργίας, η μελλοντική μορφή της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλά εδώ τώρα έχουμε μια έκθεση ως απάντηση στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 29 Νοεμβρίου και έτσι έχουμε την ουσιαστική συζήτηση ω απάντηση στην ανακοίνωση αυτή. Ασφαλώ θα σα πει περισσότερο η συζητητή ο ίδιο και για το χρονοδιάγραμμα. Και προτείνω να τον ακούσουμε αμέσως μετά θα ακούσουμε τους και οδησηγητές και τους συντονιστές ή τους αντιπροσώπους τους. Αν δέχεστε λοιπόν την ημερήσια διάταξη, παρακαλώ τον κύριο Ντόρφμαν τον να λάβει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Ε, θα συνεχίσω εκεί που σταθήκατε εσείς, το χρονοδιάγραμμα δηλαδή. Είχαμε πει ότι θα ήταν καλό αν μπορούμε μέσα στο Μάιο, το αργότερο μέσα στον Ιούνιο, να έχουμε ε, μια συνεδρίαση εδώ στο Στρασβούργο για την ε, λήψη απόφαση για την έκθεση αυτή. Αυτό σημαίνει ότι στις 17 Μαΐου μπορούμε να ψηφίσουμε, μάλλον πρέπει να ψηφίσουμε στις 17 Μαΐου στην Επιτροπή Γεωργίας. Έχουμε λίγο χρόνο, λίγο χρονικό περιθώριο, γι' αυτό και προσπάθησα ε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα να καταρτήσω αυτή την έκθεση, την έχετε λάβει. Θα τη εδώ στην Επιτροπή μας. Και βεβαίως θα συνεχιστεί σε επόμενες εβδομάδες και μήνες η δουλειά. Στόχος μου ήταν και είναι στην έκθεση αυτή να διατυπώσω όσο το δυνατόν το θέμα σε πολιτικού όρου, να είναι πολιτική έκθεση. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι καθήκον μια τέτοια έκθεση είναι να γράψει, να συντάξει μια νέα κοινή γεωργική πολιτική, ε, να υπησέλθει σε τεχνικά θέματα. Αυτό θα είναι ζήτημα τη νομοθετική πρόταση. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να μιλήσουμε για τι αρχέ. Να τοποθετηθούμε στα βασικά ζητήματα της ε, κοινή γεωργικής πολιτικής ή τουλάχιστον να επιδιώξουμε να διαμορφώσουμε μια ε, θέση της πλειοψηφία. Και γι' αυτό με αυτό το πνεύμα προσπαθώ να καταρτήσω την έκθεση καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ζητήματα αλλά σε επίπεδο όσο δυνατόν γενικό και όχι λεπτομέρειας ή τεχνικό. Τρία κεφάλαια ε, απαρτίζουν την έκθεση. τα οποία κεφάλαια πιστεύω ότι θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν ε, τα τρία τμήματα αντίστοιχα της νομοθετικής πρότασης. Ο Επίτροπος Χόγκαν άλλωστε σε μια προηγούμενη ε, συνεδρίαση είχε πει ότι σκόπευε να καταθέσει τρεις νομοθετικές προτάσεις, μία που θα φορούσε μια νέα σχέση επικουρικότητας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών και περιφερειών αντίστοιχα. Το λεγόμενο New Delivery Model, ένα νέο μοντέλο συνεργασίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών, όπως είναι γνωστό εδώ μεταξύ από την ε, ανακοίνωση. Μετά έχουμε την, τον πυρήνα της κοινή γεωργικής πολιτικής πρώτο και δεύτερο πυλώνας ως δεύτερο κεφάλαιο και το τρίτο κεφάλαιο είναι αυτό που έχει να κάνει με τις ε, ε, οργανώσεις αγοράς και βέβαια τα συμπεράσματα και τις καταληκτικές προτάσεις. Για να περάσω λοιπόν στο νέο, στη νέα αυτή σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης Κρατών Μελών, Περιφερειών και Γεωργών. Η, έκθεση, η ανακοίνωση της Επιτροπής μας δίνει μόνο ένα γενικό σημείο κίνησης για το πώς θα διαμορφωθεί αυτή η σχέση. Δεν δίνει αρκετές λεπτομέρειες, οι οποίες θα διευκρινιστούν αργότερα. Δεν μας δίνει κατευθύνση δηλαδή, που θα πάρει αυτό το μοντέλο, αυτή η νέα σχέση. Και έτσι ε, επισημαίνω ότι αυτή η σχέση, η νέα σχέση θα πρέπει να περάσει μέσα από την απλούστευση, από την ελάφρυνση του διοικητικού βάρους ε, της κοινή γεωργικής πολιτικής και να είναι ε, δυνατή η προσαρμογή στις συνθήκες των κρατών μελών. Ωστόσο σημειώνω ότι δεν μπορεί να μην είναι πλέον κοινή η γεωργική πολιτική. Θα πρέπει να παραμείνει κοινή, θα πρέπει να παραμείνει ε, κοινή γεωργική πολιτική και δεν μπορεί η επικουρικότητα να σημαίνει ότι το κάθε κράτος μέλος θα κάνει ό,τι θέλει. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα με την παραγωγή τροφίμων στη γεωργία μας, να καλύπτουμε τις δυνατότητες ε, για ε, λήψη αποφάσεων, επιτρέπουμε λέει, τη λήψη αποφάσεων από τα κράτη-μέλη με την αρχή της επικουρικότητας, χωρίς όμως αυτές να οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Επίσης αναφέρομαι σε μια γενική ε, σε ένα γενικό σχεδιασμό ή προγραμματισμό της γεωργικής πολιτικής σε επίπεδο κράτους, που προτείνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα σχεδιασμό προγράμματος λοιπόν εφαρμογή και έλεγχο στο πλαίσιο της προσέγγισης, μέσα σε ένα πυλώνα. Και αυτό το λέω διότι ε, υπάρχουν δυνατότητες σχεδιασμού ή προγραμματισμού στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε αυτά τα οποία έχουν ομοσπονδιακό χαρακτήρα. Είναι πολλαπλά τα επίπεδα του σχεδιασμού, ε, γιατί και για το πρώτο και για το δεύτερο πυλώνα μπορεί να έχουν αρμοδιότητες όχι μόνο τα κράτη σε κεντρικό επίπεδο, αλλά και οι περιφέρειες. Έτσι λοιπόν η νέα πρόταση δεν μπορεί να οδηγήσει σε αποστέρηση από τις περιφέρειες των αρμοδιοτήτων που έχουν σε σχέση με το σχεδιασμό, ιδιαίτερα του δεύτερου πυλώνα, ε, αρμοδιότητες μάλιστα οι οποίες απορρεύουν από τη σταγματική τάξη του κράτους. Δεύτερο τμήμα, δεύτερο κεφάλαιο, εκεί που γίνεται αναφορά στον πρώτο και δεύτερο πυλώνα. Εδώ σημειώνω ότι πρέπει, ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η τρέχουσα δομή των δύο πυλώνων και ο πρώτος ιδιαίτερα έχει αποδείξει την αξία του. Θα πρέπει να διατηρηθεί λοιπόν αυτή η δομή, τουλάχιστον αυτό υποστηρίζω εγώ. Και ταυτόχρονα λέω ότι θα πρέπει να, είναι, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ε, κάλυψη οικονομική. Έτσι λοιπόν η κοινή γεωργική πολιτική στο προσεχές δημοσιονομικό πλαίσιο θα πρέπει να έχει τουλάχιστον την πρικοδότηση σε όρους δημοσιονομικούς που έχει μέχρι τώρα, μέχρι το υφιστάμενο. Πού για να καλυφθούν οι φιλοδοξίες ε, με τρόπο αποτελεσματικό σε οικονομικούς όρους. Επίσης κάνω μια παρατήρηση για τον πρώτο πυλώνα, το ευρωπαϊκό αυτό μοντέλο γεωργίας, το οποίο στηρίζεται σε οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του γεωργικού προτύπου της Ευρώπης ένα, ένα μοντέλο, ένα χαρακτηριστικό το οποίο θα πρέπει να προωθήσουμε. Εδώ έχουμε να κάνουμε με οικογενειακές επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις που σε διαφορετικές περιοχές, περιφέρειες, τόπους της Ευρώπης έχουν και διαφορετικό μέγεθος και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους μηχανισμούς εκείνους οι οποίοι θα διαφυλάξουν τις μικρές και μεσέ ε, εκμεταλλεύσεις, θα τους επιτρέψουν να επιβιώσουν Έτσι λοιπόν μια σταδιακή αναλογική μάλλον σε σχέση με το μέγεθος μείωση των ε, ενισχύσεων στον πρώτο πυλώνα θα είχε λογική και μάλιστα θα αντιμετώπιζε τους κινδύνους τρευλώσεων των, ε, ε, του ανταγωνισμού. Ωστόσο, ε, το απόλυτο capping, δηλαδή το αν θα τεθεί ένα απόλυτο και ανυπέρθετο όριο στις ενισχύσεις, είναι μια απόφαση την οποία εγώ θα προτιμούσα να αφήσουμε στα κράτη. Επίση, το υπάρχον σύστημα υπολογισμού των άμεσων ενισχύσεων στην πυλώνα 1 συχνά βασίζεται σε ιστορικά δικαιώματα και έτσι θα μπορούσε σιγά σιγά, να, και πρέπει να το σκεφτούμε αυτό, θα μπορούσαμε λοιπόν να βρούμε μια λύση η οποία σταδιακά θα προχωρούσε σε ένα διαφορετικό και πιο σύγχρονο σύστημα. Έτσι το 2027 θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα βαζόταν σε ιστορικά δεδομένα του 2000, δηλαδή 27 ετών πίσω. Ένα σύστημα λοιπόν ενιαίο και πιο απλό και πιο διαφανές. Θα μπορούσε βεβαίω να αντικατασταθεί το σύστημα, των ε, άμεσων ενισχύσεων εντελώ και να αντικατασταθεί από ένα πιο απλό σύστημα. Η εσωτερική σύγκληση στα κράτη-μέλη είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να επιδιώκουμε με τη χρηματοδότηση, με τις ενισχύσεις, αλλά και στην κατανομή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το γεγονός ότι υπάρχουν διαφορετικό κόστος, παραγωγής συνθήκες παραγωγής ανάλογα με την περιοχή και περιφέρεια τη ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και μεταξύ των κρατών μελών. Δεν μπορούμε να το γνωρίσουμε αυτό. Πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν συνολικά τον πρώτο και δεύτερο πυλώνα και όλο το σύστημα χρηματοδότησης της γεωργίας. Επίσης, τι συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις δεν μπορούμε να τις εγκαταλείψουμε, τις χρειαζόμαστε ακόμα, απλώς πρέπει να μεριμνήσουμε να μην οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Στο ζήτημα των γενναιών, στην ανανέωση των γενναιών, έχουμε να κάνουμε μια μεγάλη πρόκληση. Μια εθνική στρατηγική πρέπει να επιληφθεί στα κράτη-μέλη του ζητήματο αυτού μέσα στον πρώτο πυλώνα, αλλά και με στοχευμένα μέτρα στο δεύτερο πυλώνα. Χρειάζονται χρηματοδοτικά μέσα και εθνικά μέτρα για να δοθούν κίνητρα στους γεωργούς, αλλά αυτά δεν μπορούν να εξαντλούνται στην κοινή γεωργική πολιτική. Θα πρέπει και άλλα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο που ε, θα μπορούσαν να αναφέρονται στο φορολογικό δίκαιο, σε ένα σύστημα στο εξοδοτικό, εθνικό, να δώσουν κίνητρα για την ανανέωση των γενναίων. Αναφέρομαι επίση στο, η σημασία του δεύτερου πυλώνα, το υπογραμμίζω τη σημασία τη αγροτική Ανάπτυξη και τη Πρωτοβουλία Λίντερ Ιδιαιτέρω. Ένα άλλο σημείο πολύ σημαντικό που θα μας απασχολήσει και τον ε, Απρίλιο είναι αυτό του ε, πράσινίσματος των οικολογικών δηλαδή περιβαλλοντικών ε, παρεμβάσεων, πώς μπορεί να αιτιολογηθούν δηλαδή δημόσιες παρεμβάσεις οικονομικές στο χώρο των περιβαλλοντικών, τα περιβαλλοντικά μέτρα. Εδώ πρέπει να κάνουμε πιο απλά τα πράγματα, λιγότερη γραφειοκρατία χρειάζεται. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει επαρκής έλεγχος ε, της υλοποίησης των δεσμεύσεων προς το περιβάλλον, προς τον οικολογικό προσανατολισμό. Δεν θα καταργηθεί δηλαδή το greening, δεν θα έχουμε ε, υποβάθμιση της σημασίας του οικολογικού προσανατολισμού, απλώς πιο απλά μέτρα. Σημαντική βεβαίως είναι οι διάσταση καινοτομίε για το, οι του μέλλοντος στη γεωργία μας. Αυτό πρέπει να λάβει ακόμη μεγαλύτερη σημασία στα επόμενα χρόνια. Και κλείνοντα καλό να ε, αναβαθμιστεί η αναγνώριση του ρόλου των παραγωγών στο, στην αλυσίδα των τροφίμων, είτε πρόκειται για ε, το τομέα, τρόφιμα και άλλους διάφορους τομείς της γεωργικής παραγωγής. Χρειαζόμαστε μέτρα ενίσχυσης του ρόλου και της, παρου... αναγνώρισης του ρόλου αυτού στην αλυσίδα τροφίμων. Η αγορά του γάλακτος επίσης έχει κεντρική σημασία εδώ και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει και πάλι το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε, να υποστηρίξουμε εθελοντικές ε, συνεργασίες και συμπράξεις στον χώρο του γάλακτος. Γιατί ακόμα αυτό δεν έχει εξασφαλιστεί. Δεν έχει ε, μηχανισμοί κρίσεως. Πρέπει και αυτοί να βελτιωθούν. Έστω και μέσα από την κατάργηση του χαρακτήρα του ενιάυσου προϋπολογισμού. Ίσως θα έπρεπε να καταργηθεί αυτό για να εξασφαλιστεί ένα ταμείο πιο ογκώδες το οποίο θα μας επιτρέπει στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσεις όποτε αυτές εμφανίζονται. Σημαντικές επίσης είναι οι ε, εμπορικές συμφωνίες. Είναι πολύ σημαντικές, πρέπει όμως να είναι και δικές και να μην ανοίγουν την αγορά σε προϊόντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τη γεωργία. Ολοκληρώνοντας, ε, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε ταχαίως τις εργασίες μας. Τον Ιούνιο, όπως είπαμε, θα έχουμε την νομοθετική πρόταση και άρα ε, λιγότερο από 12 μήνες πριν από το πέρας της θητείας ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη δουλειά. Ε, μακάρι να είχαμε τα κείμενα νωρίτερα και να μπορούσαμε να κάνουμε με πιο πολύ περιθώριο χρονικό αυτή τη δουλειά εκ μέρου του Κοινοβουλίου. Πρόεδρε, αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της ε, έκθεσής μου. Σας ευχαριστώ όλους όσοι με βοήθησαν ιδιαίτερα τις τελευταίες εβδομάδες, με στήριξαν, μου έδωσαν ιδέες, ε, με όθησαν να ολοκληρώσω την έκθεση, τους σκιώδεις ηγητές ιδιαίτερως, αλλά και το προσωπικό μας, τη γραμματεία μας που ε, συνέβαλε τα μάλα σε αυτή τη δουλειά και ελπίζω αυτή η συνεργασία με τους συναδέλφους να συνεχιστεί και στη φάση των τροπολογιών. Θα προχωρήσουμε στο μέγιστο δυνατό να συμπεριλάβουμε τις τροπολογίες μέσα στο κείμενο και για να ολοκληρώσω θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους να δεχθούν τη βασική αρχή ότι δεν πρέπει να ε, παρασυρθούμε σε τεχνικές ε, λεπτομέρειες, σε μεγάλο βαθμό ε, λεπτομέρειας, αλλά ότι θα πρέπει να περιοριστούμε στην ανάπτυξη γενικών αρχών και να αφήσουμε το τεχνικό ζήτημα, τις τεχνικές λεπτομέρειες, στη δουλειά που θα ακολουθήσει ο επόμενος μήνες, που είναι οι νομοθετικές προτάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Κύριο ο συγητής θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει στο τέλος της συζήτησης. Έχουμε 30 ομιλητές στον κατάλογό μου. Σκιώδης συζητητές με τα συντονιστές. Δύο λεπτά για τον καθένα. Και μετά ένα λεπτό για κάθε ε, βουλευτή κυρία Αγγιλέρα. Παρακαλώ, θα σας ειδοποιώ 10 δευτερόλεπτα πριν να ε, λήξει ο χρόνος σας. Οπότε έχετε, ε, κοιτάτε με ώστε να γνωρίζετε πότε πρέπει να τελειώσετε. Η κυρία Γιλαρά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ναι, με προειδοποιήσατε, κατάλαβα με το σφυράκι σας. Είναι αλήθεια ότι συμβαίνει το εξής. Για πρώτη φορά συγκροτείται σήμερα η Ειδική Επιτροπή για τα φυτοφάρμακα. Οπότε τα τελευταία 45 λεπτά θα πρέπει να φύγω και δεν θα ακούσω την ε, δευτερολογία του εισηγητή. Δεν θα αναφερθώ σε όλες τις στοιχείες της έκθεσης και θα επικεντρωθώ σε κάποια επιμέρους σημαντικά ζητήματα. Να τον ευχαριστήσω καταρχάς για τη δουλειά του και για το ότι μας έδωσε αρκετό χρόνο για να προσεγγίσουμε ένα θέμα με αρκετό χρόνο για συζήτηση και για τροπολογίες. Εγώ να τονίσω το εξής. Δεν επισήλθαμε σε λεπτομέρειες τεχνικές. Εδώ χαράζουμε πολιτικές κατευθυντήρες γραμμές για τις οποίες για κάποιες συμφωνώ, για άλλες διαφωνώ. Πάντως αυτές οι κατευθυντές γραμμές πρέπει να είναι ξεκάθαρες, δηλαδή δεν θα πρέπει να έχουμε επαναθνικοποίηση, δεν θα πρέπει να έχουμε συγχρηματοδότηση, όμως στην ανακοίνωση αυτά θα πρέπει να είναι σαφή και να μην υπάρχουν αμφιβολίες σε σχέση με αυτά. Γιατί προσωπικά θεωρώ περίπλοκη όλη αυτή τη ε, διαδικασία όπου είναι εύκολο να γίνουν προσαρμογές σε ένα πυλώνα ε, και να υπάρχει χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον άλλο πυλώνα να υπάρχει συγχρηματοδότηση. Εγώ λοιπόν έχω πολλές αμφιβολίες σε σχέση με τη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε. Παρόλο που για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων συμφωνώ. Να τονίσω και κάτι άλλο. Η πράσινη δομή, η πράσινη αρχιτεκτονική θα πρέπει να είναι ξεκάθαρη στην ανακαίνωση. Δηλαδή, ποιο είναι το πρότυπο που θα πρέπει να υπερισχύσει στην Ευρώπη. Επίσης, η κοινή γεωργική πολιτική θα πρέπει να επαφείται στις χώρες μέλη. Θα πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη ασφάλεια όταν θα καθορίσουμε ευρωπαϊκούς κανόνες για την κοινή γεωργική πολιτική. Και κατά λίγο, Πρόεδρε, για τα θέματα διαχείρισης κρίσεων. Θα πρέπει να βελτιωθεί κατά πολύ αυτό το ζήτημα και απέχει πολύ από το να αριθμιστεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, και Πρόεδρος. Πάντω ε, θα ήθελα να σα ε, ζητήσω, λέει ο Πρόεδρο, να μην σπατάσουμε χρόνο στι ευχαριστίε και να μιλήσουμε για τα πιο σημαντικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Ο Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να πω και εγώ καταρχά ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε γιατί δαπάνησε χρόνο και δύναμη για αυτό το τόσο συνεκτικό έγγραφο. Εγώ τα έχω ξανά αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε για μεταρρυθμίσει της ΚΑΠΑΓΑΜΑΠ είχαμε το θέμα του προπολογισμού και ο εισηγητή το ξέρει καλά αυτό. Δηλαδή όλοι θέλουν να αποσπάσουν τμήματα από το δικό μας προπολογισμό για να επεκτείνουν, να διευρύνουν τέλο πάντων τα δικά τους τα θέματα, όπως νομίζουν. Και νομίζω ότι αυτό επιβαρύνεται και από την αναχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου και τη συμμετοχή του στον προπολογισμό. Δεν ξέρω κατά πόσο πρέπει να χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά δυστυχώ έτσι έχουν τα πράγματα. Πάντω, αυτό ενσυχεί του εμπλεκόμενου στη Γεωργία και το θέμα νομίζω πηγαίνει πέραν τη τωρινή θητεία του Κοινοβουλίου. Εγώ ίσω να μην είμαι στην επόμενη βέβαια, αλλά για αυτού που θα είναι εδώ θα πρέπει να πρασπιστούν τον προπολογισμό τη κοινή γεωρικής πολιτική. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν δεν έχουμε το δέοντα προπολογισμό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί έχουμε πολλέ αβεβαιότητε, πολλά προβλήματα και δεν μπορούμε να πετύχουμε τίποτα αν υπάρχουν τα απαραίτητα κονδύλια. Και βεβαίω καλωσορίζω την εστίαση στην καινοτομία και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ καλό εκ της Κομισιόν. Θα πρέπει επίσης να δούμε κατά πόσο οι χώρες μέλη θα μπορούσαν να το, να το συμπληρώσουν αυτό με το gold plating και με τρόπο ώστε να γνωρίζουμε ακριβώς τι προσδοκάμε από τις χώρες μέλη στα θέματα αυτά. Θα πρέπει και οι πυλώνες επίσης να είναι συμπληρωματικοί, να μην αφήνουν να Νομίζω ότι ο ένας πυλώνας αυτή τη στιγμή είναι αρκετά περίπλοκος και θα πρέπει να το ρυθμίσουμε αυτό. Αυτά είχα εγώ να πω πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωραία. Και πάλι να σας παρακαλέσω. Μην ευχαριστείτε τους πάντες γιατί χάνουμε χρόνο. Κυρία Θέλω να ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν. Είναι πολύ πλήρης η έκθεση με σαφή δομή. Αναφέρεται και στην, ε, στο στόχο της απλούστευσης στη γεωργική πολιτική. Βεβαίως και μπορούμε να το υποστηρίξουμε αυτό. Ε, βεβαίως θέλουμε την απλούστευση ως το δυνατόν λιγότερους κανόνες για τον τρόπο που θα έχει κανείς στην εργασία του στον χώρο της γεωργίας για τον, ε, για τον προϋπολογισμό θα συμφωνήσω με τις ανησυχίες του συναδέλφου κυρίου Νίκολσον γιατί δεν ξέρω αν είναι δυνατόν να διατηρηθεί αυτός ο προϋπολογισμός για τις εκμεταλλεύσεις. Αναφέρεται σε μικρότερες εκμεταλλεύσεις ε, ο κύριος Τόρφαμαν, αλλά θα ήθελα να συμπεριλάβει και τις μεσαίες εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο δεν βλέπω επίσης θέματα βιοοικονομίας και δασοπονίας, ίσως κάπου στο σημείο 16, εκεί που γίνεται λόγος και για τον αγροτουρισμό θα μπορούσαμε να τα συμπεριλάβουμε. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τα Πρωτοενούχα επίσης ε, με ανησυχεί στο δεύτερο πυλώνα. Η Γερμανία είναι η μόνη η οποία δεν έχει συνδεμένες ε, ε, ενισχύσει και αν δούμε τα όσα αναφέρονται στον κανονισμό Omnibus δεν θα έπρεπε να υποστηρίζουμε περαιτέρω την ε, καλλιέργεια πρωτεϊνούχων. Θα ήταν καλό λοιπόν να συνδεθούν εδώ οι ενισχύσεις. Αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, βεβαίως, στο πλαίσιο του κανονισμού Omnibus έχουμε εξασφαλίσει πολλά, πολλές λύσεις ε, βασικές αποφάσεις που έχουν βεβαίως να κάνουν και με τη διάθεση των κονδυλίων, μια φάση μεταβατική δηλαδή μέχρι την ε, θέση εφαρμογή της νέας κοινή γεωργικής πολιτικής πρέπει να εξασφαλιστεί. Είναι σημαντικό αυτό, χρειάζονται λοιπόν μεταβατικές διατάξεις. Εν όλο, στην κοινή οργάνωση αγοράς νομίζω ότι καλύπτονται σε σχέση με αυτά που έχουμε αποφασίσει και βεβαίως θα καταθέσουμε τις τροπολογίες αναλόγως ε, στα θέματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν συνεχίσουμε με την ίδια κάμπα γάμα πι, θα συνεχίσουμε να παραπονιούμαστε μετά από πέντε χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να διαφυλάξουμε τα εισοδήματα των γεωργών. Εδώ ακούμε μόνο δηλώσει προθέσεων και δεν γίνεται καθόλου λόγος για τα δικαιώματα των γεωργών. Δεν είδαμε να υπάρχουν επίσης συγκεκριμένες λύσει που να αφορούν το θέμα της ε, μεταβολής των τιμών. Και νομίζω ότι οι διάφορες τομιακέ συμφωνίε που έχουμε γίνονται σε εθελοντική βάση και είδαμε ότι αυτό ακριβώς απέτυχε στον τομέα των γαλακτοκομικών. Θεωρώ λοιπόν θα πρέπει η πρότασή μας να είναι πολύ πιο φιλόδοξη η οποία θα διασφαλίζει το ότι στο μέλλον θα έχουμε γεωργούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι οποίοι θα μπορούν να επιβιώσουν στις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αναφέρθηκε ήδη. Θα προεκριθούν τα πάντα από το πώ θα διαμορφωθεί ο προπολογισμό μα στην επόμενη δημοσιονομική περίοδο. Εάν δεν μπορούμε να πούμε ξεκάθαρα πώ μπορεί να συμβάλλει η γεωργία στην καταπολέμηση τη κλιματική αλλαγή, πώ στηρίζει τη βιοπικιλότητα, πώ εξασφαλίζει τη διατήρηση τη συνεργασία, τότε θα είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθεί αυτό ο προπολογισμό που είχαμε μέχρι τώρα. Αυτό που δεν βλέπω εγώ στην έκθεση είναι αναφορά σε, στην Ήπεθρο σε, σε περισσότερα σημεία της έκθεσης. Πρέπει περισσότερο να τονιστεί ο ρόλος της Ήπεθρου, πόσο συμβάλλει, πώς αξιοποιεί τα χρήματα, τι, τι, τι ωφέλη προσφέρει. Επίσης, την παράγραφο 25, εγώ δεν συμφωνώ, διότι θεωρώ ότι πρέπει κατά κύριο λόγο χρήματα του Ευρωπαίου ε, φορολογούμενου να αξιοποιούνται για την αυτονομία και την ε, πρώτο καθεδρία, την διατροφική της Ευρώπης και όχι για να παίζουμε μέσα στις παγκόσμιες αγορές εμπορίου. Αντιστρόφως, τρόφιμα τα οποία εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υφίστανται, να ε, υπόκεινται στις ίδιες ε, προδιαγραφές με τις προδιαγραφέ που ισχύουν για τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Παραδείγματι, έχουμε ένα θέμα με τι εισαγωγέ ε, αυγών ε, από συστοιχίε, παραγωγή σε συστοιχίε. Ε, ένα άλλο θέμα είναι η χρήση χρημάτων των φορολογουμένων για την ανάπτυξη δυτικού κέρδους. Και εδώ δεν μπορώ να συμφωνήσω βεβαίως. Ή τα ποσά τα οποία πηγαίνουν στην περιβαλλοντική υποστήριξη, τη βιοποικιλότητα. Εδώ θα ήθελα να υπάρχει μια υποχρεωτική ελάχιστη, ένα ελάχιστο ποσοστό. Κάτι άλλο το οποίο δεν βλέπω είναι η υποστήριξη απευθείας στην διάθεση στον καταναλωτή, την ε, επιχείρηση, την αγροτουριστική κτλ. των προϊόντων. Αυτό θα έχει νομίζω μεγάλη σημασία να το υποστηρίξουμε μαζί με την ανάπτυξη μιας ε, αγοράς ε, η οποία θα στηρίζει τον ε, γεωργό. Η δε σταδιακή και αναλογική μείωση ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης των ενισχύσεων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική και ραγδαία. Το κάπινγκ λοιπόν πρέπει και επειδή ε, παρουσιάζεται σημαντικό κίνδυνος ανταγων, ε, στρέβλος του ανταγωνισμού να έχει την ίδια, ε, την ίδια κάλυψη. Ναι, το κλείνω κύριε Άντνιου, το κλείνω. Ευχαριστώ. Η εκθέση του συναδέλφου μου φαίνεται ότι έχει απόλυτη ισορροπία αλλά θέλω λίγο να αφισβητήσουμε τι πολιτικέ αρχέ, Να δούμε λίγο τι πολιτικέ αρχέ συγγνώμη, που πρέπει να διασφαλίζει αυτή η έκθεση. Κάτι ανησυχητικό πρώτα απ' όλα είναι αυτό το νέο μοντέλο παράδοση, το New Delivery Model, το οποίο παρά ε, τις διαβεβαιώσεις της Επιτροπής ενέχει τον κίνδυνο εκ νέου ε, ε, εθνικοποίησης κατά κάποιο τρόπο της ΚΑΠ, δηλαδή το να δοθεί στα κράτη-μέλη υπερβολικός έλεγχος ε, της εδαφικής πολιτικής. Πέραν ε, δηλαδή από κάτι το οποίο θα έπρεπε κανονικά να είναι κοινό στόχο. Όταν μιλάμε λοιπόν για κοινή γεωργική πολιτική, ε, χρειάζεται κάποια διαχείριση, κάποιοι στόχοι κοινοί. Θα πρέπει να καταπνίξουμε τη γενέση τους μηχανισμούς που αναφεθούν ε, στην ε, ελεύθερο ανταγωνισμό της αγοράς μπορεί να οδηγήσουν σε ανταγωνιστικές ε, δυναμικές αθέμητες τιμωρώντας έτσι ολόκληρο τον τομέα. Πρέπει να δοθεί λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή στην έννοια της εξωτερικής σύγκλησης. Και σε αυτή την περίπτωση, όταν μιλάμε για κοινή πολιτική, δεν μπορούμε να μην λαμβάνουμε υπόψη ποιο είναι το κόστος ζωής και εργασίας στα διάφορα κράτη-μέλη και σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην ε, δημιουργήσουμε υπερβολικές πολιτικές αθέμη του ανταγωνισμού. Στο άλλο μέτωπο, συνεπώς, ε, είναι κατά την άποψή μα απαραίτητο να εισάγουμε μηχανισμούς ε, επιβράβευσης, δηλαδή να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που συμβάλλουν θετικά στο περιβάλλον κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά. Που ακολουθούν δηλαδή κάποια προοδευτική προσέγγιση όσον αφορά τις στηρίξεις και που βοηθάν να καταπολεμηθούν όλοι οι μηχανισμοί αρπαγής γης που δημιουργούν τόση βλάβη στον τομέα. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση που ακολουθεί ε, την ανακοίνωση της ε, Κομισιόν ανακοινώνει τη συζήτηση 2020-2027 ε, ε, ε, για την ΚΑΠ για αυτή την περίοδο. Θα πρέπει να φοβόμαστε ότι μπορεί να μην υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος της θητείας του Κοινοβουλίου. Αυτό φοβάμαι ότι μειώνει το χρόνο που έχουμε για να συζητήσουμε και τελικά οι επιθυμίες της Κομισιόν θα περάσουν στις ανταλλαγές μας λοιπόν θα πρέπει να υπερασπιστούμε τους γεωργούς και τη γεωργία στα κράτη μας. Αυτό το κείμενο λοιπόν δείχνει ε, υπό τα σημεία 1, 2 και 3 ότι δεν υπάρχει καμία βούληση να δοθεί ελεύθερη επιλογή στα κράτη-μέλη, προωθείται η κοινή αγορά, η ενιαία αγορά, περιορίζεται η ευελιξία που έχουν τα κράτη-μέλη για να ορίσουν κάποιου κανόνε, ε, δεν λαμβάνεται υπόψη η επικουρικότητα. Δεν συμφωνούμε απόλυτα. Θεωρούμε και εγώ ω Γάλλο Γεωργό ότι αυτά δεν είναι σωστά. Στο σημείο 9 είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέγεται. Πρέπει να διατηρηθεί ο προπολογισμό. Στο 10 ε, το 10 αντιβαίνει ε, στις συνέπειες της ΚΑΠ μετά από δεκαετίες όπου συχνά η ΚΑΠ ε, είναι μια υπερφιλελεύθερη ε, πολιτική και ε, έχει επηρεάσει αρνητικά πάρα πολλέ επιχειρήσει στη Γαλλία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν λαμβάνεται υπόψη η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου που αναφέρεται στην αναποτελεσματικότητα τη πολιτική όσον αφορά την ανάπτυξη τη υπαίθρου. Εγώ μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι είναι αποτυχία και αποτελεί η μεταρρύθμιση των ε, ε, μειονεκτησών περιοχών ε, μια απόδειξη. Το 25 είναι ένα θετικό σημείο, είναι μια αρχή όπου αναγνωρίζεται ότι κάποιες δυσκολίες οφείλονται στις εμπορικές συμφωνίες και αυτό απαιτεί παγίαση των μηχανισμών διασφάλισης για να υπάρχει θεμητός ανταγωνισμός. Θέλω μια νέα κάπα που να προσφέρει επισητιστική ασφάλεια αναπτύσσοντας τις αλυσίδες με γεωργικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να είναι προσοδοφόρο για τους γεωργούς και να εξυπηρετεί η ΚΑΠ αυτή τους γεωργούς αντίθετα από το δεύτερο κεφάλαιο το οποίο έχετε ξεχάσει κύριε Ισηγητά. Τέλος, θεωρώ ότι αυτή η ΚΑΠ στο επίκεντρο των αποφάσεων πρέπει να θέτει το γεωργό και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο. Θα πρέπει να επιμένουμε σε αυτό. Ο Ευχαριστώ. Η έκθεση υπενθυμίζει ότι η κοινή γεωργική πολιτική ε, υποστηρίζει τα ε, εισοδήματα των γεωργών. Είναι μια στήριξη σε έναν οικονομικό τομέα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Το γεγονός ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα στρατηγική δεν πρέπει να μας κάνει να ξεχνάμε ότι το σύστημα αιρεσιμότητας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι μια κοινή βάση για όλους τους Ευρωπαίους γεωργούς. Δεν πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ της υλοποίησης ε, στις διάφορε χώρε. Διαφορετικά αυτό δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ μας. Πρέπει να διατηρήσουμε την ακυρεότητα του πυλώνα 1, περιορίζοντας ε, στο 30% ε, τις, τις συμμετοχές. Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστές από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμή με το greening θα πρέπει να συμφιλιώσουμε την οικονομία και το πρασίνισμα. Για οποιαδήποτε μορφή γεωργία και αν μιλάμε, είτε μιλάμε για γεωργία διατήρηση, ευφυή, γεωργία κτλ. Σε όλα αυτά τα προγράμματα έχουν δεσμευτεί οι γεωργοί, είναι ενάρετα προγράμματα και η ΚΑΠ θα πρέπει να τα αναγνωρίσει. Ο δεύτερο πυλώνα τη ΚΑΠ θα πρέπει να συμπληρώνει τι επενδύσει που είναι απαραίτητε στον πρώτο πυλώνα για την ανάπτυξη. Αυτό πρέπει να κάνουμε για παράδειγμα στη γεωργία ακριβία. Επίσης, στο επίπεδο της οργάνωσης των αλυσίδων, οι συνδεδεμένες ε, ενισχύσεις έχουν ε, βοηθήσει και είναι αποτελεσματικές, αλλά έχουν όρια. Το, πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα στον τομέα των φρούτων και λαχανικών θα πρέπει να μας βοηθήσει να προωθήσουμε και άλλους τομείς οικονομικά. Τέλος, δεν μπορεί να υπάρχει ΚΑΠ χωρίς ένα πραγματικό αποθεματικό για περίοδους κρίσης. Θα πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε αυτό το επαθηματικό για να γίνει πραγματικά λειτουργικό. Ο κύριος Αντρίου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πραγματι θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου πέρα από την έκθεση του συναδέλφου που είναι ποιοτική και να μιλήσουμε για τα οικονομικά ζητήματα και να διασφαλίσουμε δηλαδή την οικονομία της γεωργίας και των γεωργών Νομίζω ότι αυτές οι προτάσεις θα πρέπει να τις εμβαθύνουμε. Γιατί καμιά φορά ξεχνάμε ακριβώς την αστάθεια που υπάρχει στις τιμές, που είναι το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στη Γεωργία και θα πρέπει να προβλέψουμε κάτι όταν δεν λειτουργεί σωστά η αγορά. Νομίζω ότι θα πρέπει ε, να υπάρχει η σωστή λειτουργία του συστήματος των εγγύησεων. Θα πρέπει λοιπόν να κινητοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και θα μπορούσαμε να προβλέψουμε και ένα απόθεμα, ένα αποθεματικό κρίσης και να έχουμε αυτή τη δυνατότητα σε επίπεδο πολιετές ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αν συμβεί κάτι θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το αποθεματικό κρίσης για να ρυθμίσουμε ακριβώς τα προβλήματα αυτού του τομέα. Θα πρέπει να αλλάξουμε τις αγορές, αυτό είναι απαραίτητο, αν θέλουμε πραγματικά να καταλήξουμε στην ολοκλήρωση αυτών των μετατροπών, ώστε να λαμβάνουν να αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους και να εξοκινεύουν περισσότερο οι γεωργοί. Μετά, για τα πρότυπα εφαρμογής. Νομίζω θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να έχουμε κατά νου τους στόχους. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι η Κομισιόν μιλάει πούμε, για τις εθνικές δεσμεύσεις και δεν μιλάει για τις λειτουργικές δεσμεύσεις. Και σε επίπεδο εργαλείων και σε επίπεδο δράσεων η διάσταση είναι πανευρωπαϊκή, ανεξάρτητα από τους στόχους. Και τέλος υπάρχει κάτι άλλο το οποίο θα πρέπει να μας ανησυχήσει. Για τους σπόρους υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να πάμε να εντάξουμε μάλλον περισσότερους γεωργούς προς το κοινό συμφέρον της γεωργίας και της κοινωνίας. Ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, ο ομιλητής. Νομίζω ότι η μεταβατική φάση του Brexit θα μπορούσε να κρατήσει επάπειρον. Οπότε το ίδιο και οι συζητήσεις για αυτά τα θέματα στη Βρετανία. Εγώ ανησυχώ για αυτό τον όρο οικογενειακές εκμεταλλεύσεις Είναι κάτι υποκειμενικό, δεν σημαίνει κάτι. Οι Κομισιόν αναμένουμε να υποβάλουν ένα σωστό προσχέδιο, αλλά πώς θα προσδιορίσουν ακριβώς τον όρο οικογενειακή εκμετάλλευση. Αν το αφήσουν αυτό να το προσδιορίσουν οι χώρες μέλη, τότε εντάξει. Αν έχουμε πληρωμές από τον πρώτο πυλώνα, τότε θα έχουμε λήψει στο δεύτερο πυλώνα. Και είχαμε πρόσφατα σε μία επιτροπή εδώ στο Κοινοβούλιο, προπολογισμό, έχω προπολογισμό, δεν θυμάμαι, κάποιο έλεγε από την Κομισιόν ότι μόνο, τα, μόνο το 50% των χρημάτων των κοντιλίων του δευτέρου πυλώνα δίδονται επειδή η διαδικασία είναι πολύ περίπλοκη. Αν λοιπόν έχουμε λήψει στον δεύτερο πυλώνα και τα χρήματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τα κονδύλια δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν, τότε χάνουμε όλοι. Ένα άνθρωπο από το Κόμμα των Πρασίνων μίλησε για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Πρόσφατα, επιστήμονε από Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΕΙΠΑ, χρησιμοποιώντας ε, τεχνολογία ε, κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν για συγκεκριμένα, συγκεκριμένες καλλιέργειες φυτών μόνο το 75% του νερού που χρειάζεται. Έχετε λοιπόν απαντήσεις. Ε, οι απαντήσεις αυτές δεν προχωρούν από την Αυστρία, τη Γερμανία, αλλά από άλλες χώρες και άλλους επιστήμονες. Τι θα κάνετε λοιπόν, θα τις απορρίψετε αυτές τις νέες τεχνολογίες ή θα τις αποδεχτείτε. Ευχαριστώ. Κύριος Χόισλινγκ, ναι, να οργανώσουμε μια βρετανική πολιτική και όχι ευρωπαϊκή για να μπορεί να μιλάει ο κύριος Άγνιο εγώ θεωρώ ότι είναι μια σαφή τοποθέτηση αυτή η έκθεση σε σχέση με τα όσα μας λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της που είναι η επανεθνικοποίηση ουσιαστικά. Δεν έχει τίποτε να κάνει με λιτότητα αυτή η πρόταση αλλά με επανεθνικοποίηση και σε αυτό πρέπει να τοποθετηθούμε. Ε, το τι θέλουμε με τη γεωργική πολιτική. Βεβαίως θα πρέπει να βρούμε πιο σαφείς διατυπώσεις για την υποστήριξη της ε, περιβαλλοντικής προσέγγισης δεν το καταφέραμε, δεν καταφέραμε ούτε με τη βιοποικιλότητα ούτε με την κοινή πολιτική να βελτιώσουμε την ε, κατάσταση του περιβάλλοντος. Άρα λοιπόν πρέπει να περάσουμε σε μια λογική κινήτρων με τις ενισχύσεις, δηλαδή με τις ενισχύσεις να μπορεί να κερδίσει κάτι ο Γεωργός εάν έχει μια προσέγγιση οικολογική για να του δώσουμε κίνητρα. Για το κάπινγκ δεν ε, μπορεί να ανοίξει ουσιαστικά συζήτηση γιατί αμέσως αντιδρούν ε, τα κράτη-μέλη. Ε, αλλά για τον κύριο Ντόρφμαν, αν μου επιτρέπει, θα ήθελα μία παρατήρηση. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κάποια πρωτοβουλία για το εκδομέα του γάλακτος. Ξεχάστε το, δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσετε από αυτόν επίτροπο, από τον τρέχοντα επίτροπο μέτρα. Είναι σε τελείως διαφορετικό τρυπάκι ο κύριος Χόγκαν και γι' αυτό θα ήταν καλύτερο να τα αφήσουμε αυτό. Όσως, ίσως θα ήταν όμως καλύτερο να μιλούμε για μια ε, να μιλάμε αποκλειστικά για την κυριαρχική πολιτική και όχι για τη δυνατότητα κατάκτησης των διεθνών αγορών ή για εξαγωγική στρατηγική. Επίσης, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Θα υπάρχουν συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου και στα γεωργικά προϊόντα, εάν τις θέλουμε. Ιδάλλως πρέπει να πούμε ότι δεν τις θέλουμε. Στις συνδεδεμένες ενισχύσεις και για τα πρωτεϊνούχα και για τα ε, σκάφη, τα αλλιευτικά, πάλι νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τους στόχους ε, με αυτά το, αυτό το σύστημα. Για την ε, στοχευμένη ε, στήριξη για τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Συμφωνώ αρκεί να ορίσουμε τις ε, οικογενειακές επιχειρήσεις. Οι στηρίξεις πρέπει να συνάδουν με τους στόχους της ΚΑΠ, την ενίσχυση της απασχόλησης και όσους εργάζονται αποτελεσματικά στις εκμεταλλεύσεις, στους ε, ενεργούς γεωργούς και πρέπει πραγματικά να καταλήψουμε τις ιστορικές αναφορές και θα πρέπει να ενισχύσουμε τη βοήθεια στις περιοχές με φυσικά φυσικές δυσκολίες και να ενθαρρύνουμε τις στρατηγικές παραγωγές και επίσης ε, φυσικά θα πρέπει να θέσουμε ανώτατα όρια, κάπινγκ όπω λέμε. Οι Ευρωπαίοι πολίτε σοκάρονται μερικέ φορέ επειδή οι ενισχύσει είναι υπερβολικέ. Μα ζητούν περισσότερη ταυτόχρονα όμω υποστήριξη στον γεωργικό κόσμο. Επίση θα πρέπει να δούμε το ζήτημα τη ε, με... μετανάστευση ε, όπου θέλουμε να ενθαρρύνουμε τι καλλιεργητικέ ζωέ στι χώρε και τι σχέσει του με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω και εγώ, μια και είναι και λίγος ο χρόνος, να αναφερθώ σε κάποια βασικά θέματα. Ε, δεν είναι ε, αυτός σκοπός η προάσπιση του χρήματος, αλλά πρέπει να εξυπηρετεί κάποιους στόχους το χρήμα όπως αυτό διατίθεται. Ε, χρειάζονται λοιπόν σαφείς στόχοι. Πολύ καλά όλα αυτά που μας λέτε, αλλά χρειαζόμαστε σαφείς στόχους. Δεύτερον, η αποτελεσματικότητα των κονδυλίων που έχουν μέχρι τώρα χρησιμοποιηθεί ε, έχει αποδειχθεί από ακροάσεις πολύ που έχουμε κάνει ότι δεν είναι οι απαιτούμενοι και ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιοι γεωργοί που έχουν λάβει πάρα πολύ χρηματοδότηση και έχουν προστατευτεί έναντι κάποιου ανταγωνισμού στον οποίο θα έπρεπε να είναι εκτεθειμένο, κάποιοι άλλοι έχουν πάρει πολύ λίγα χρήματα. Διαφάνεια. Διαφάνεια δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Οι ιστορικέ αναφορέ είναι δύσκολο να γίνουν κατανοητέ, να διαβαστούν και είναι και δύσκολο γιατί θα πρέπει βάσει αυτό να παίρνει κανεί χρήματα. Το σημαντικότερο για μένα ε, ερώτημα όμω είναι το πώ θα εξασφαλίσουμε την αιρεσιμότητα. Δεν είναι δυνατόν να φεύγουν αυτές οι λύσεις από τον πρώτο πυλώνα. Πρέπει να αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα της δουλειάς του Γεωργού και έτσι να τον τιμάμε, να τον ε, επιβραβεύουμε με πλήρες ως και πως όχι, το, το μισό ή το ένα τρίτο κτλ. Αλλά πρέπει εδώ να προσέξουμε ιδιαίτερα την αιρεσιμότητα στον πρώτο τιμώνα, πυλώνα. Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα και 100% αιρεσιμότητα, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος τομέας στον οποίο παίρνει κανείς χρήματα με βάση την έκταση που κατέχει. Ε, φανταστείτε να λέγαμε έφνησε ότι στην οικογενειακή πολιτική δίνουμε οικογενειακό επίπεδο ανάλογα με το μέγεθος του δωματίου του κάθε παιδιού που έχει μια οικογένεια. Θα μας ήταν Ε, αυτό προσπαθείτε να μας πείτε εδώ πέρα. Παρακαλώ. Πάνι πόσο πέτοιμη. Hvala gospodine predsjedniče, pohvaljujem nacrt izvješća koji je predložio gospodin Dorfman. Evo paraboli, to mi se gdje, ja ti nekto si Βεβαίω θεωρούμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Και αυτό νομίζω θα τα καταφέρουμε αν καλύψουμε κάποια να μέχρι την οριστική έκδοση του εγγράφου. Στην Κροατία τα εισοδήματα των γεωργών είναι χαμηλότερα από αυτά σε άλλους τομείς της οικονομίας, το οποίο σημαίνει ότι δεν προσελκύει η γεωργία νέους εργαζόμενους, νέους γεωργούς. Έχουμε λοιπόν ένα χάσμα και μια απώλεια γενεών στη γεωργία στην Κροατία. Και αυτό κυρίως οφείλεται ακριβώς στην διαφορά των εισοδημάτων. Πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους γεωργούς ιδιαίτερα να τους βοηθήσουμε και να διασφαλίσουμε την πρόσβαση σε κεφάλαια που θα τους βοηθήσουν να άρουμε φραγμούς και αποκλεισμούς και να τους βοηθήσουμε ώστε να επιδοθούν στην βιολογική γεωργία κυρίως. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο μελλοντικό προπολογισμό θα διδερματίσει σημαντικό ρόλο στην όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν πρέπει να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ενιαία αγορά και η ΚΑΠ να παραμείνει όπως έχει. Και εμείς φυσικά είμαστε κατά της εκ νέου εθνικοποίησης. Η εξωτερική σύγκληση είναι ένα επίκαιρο ζήτημα. Και όταν μιλάμε για το κάπινγκ, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την εμπειρία μας με από τα πανευρωπαϊκά μέτρα. Για παράδειγμα, όταν προσπαθούμε να ορίσουμε τους ενεργούς γεωργούς, το έχουμε ήδη κάνει αυτό και στην Omnibus τώρα λέμε ότι αναπόκειται στα κράτη-μέλη ο ορισμός. Όσον αφορά το κάπινγκ, πιστεύω ότι καλό θα ήταν να το αφήσουμε στα κράτη-μέλη, να αποφασίζουν αυτά τα ανώτατα όρια. Τώρα, ο πρώτος πυλώνας ε, και η εθελοντική συνδεδεμένη ε, στη ενίσχυση, στήριξη. Όταν μιλάμε για μικρούς και μεσαίους ε, γεωργούς, είναι σαφές ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους μικρομεσαίους, ε, μικρομεσαίου μεγέθους αγρότες. Και οι αποφάσεις μας θα πρέπει να βασίζονται όχι μόνο σε στατιστικά στοιχεία, πρέπει επίσης να λαμβάνουμε υπόψη και κοινωνικούς και πολιτικούς παράγοντες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δικαστρό. Ευχαριστώ. Η ευελιξία και επικουρικότητα είναι όμορφα λόγια, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, να μεταμορφωθούν σε μια εκ νέου εθνικοποίηση της ΠΑΚ. Της ΚΑΠ, συγγνώμη. Και όπως είπαν πολλοί ε, συνάδελφοι, δεν το θέλουμε. Ο κύριος Έμπερτ έχει, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά και πρέπει να την ενισχύσουμε. Καθαρά να πούμε ότι αυτή η Επιτροπή ουδέποτε πρόκειται να δεχθεί το New Delivery Model να μεταμορφωθεί σε μια λευκή επιταγή για τα κράτη-μέλη. Έτσι λοιπόν ε, η κίνδυνη της ε, συγχρηματοδότησης, της οικονομικής ε, διόρθωσης, της μέγιστης τρέβλωσης του ανταγωνισμού, διότι συχνά ευελιξία μεταφράζεται σε τέτοια φαινόμενα. Ήθελα να υπογραμμίσω στην ομιλία μου ένα πράγμα, όπως είπε ο συνάδελφος Ντόρφμαν. Η νομοθετική πρόταση που θα παρουσιαστεί τέλη Μαΐου από τον Επίτροπο εδώ στο Κοινοβούλιο δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να ολοκληρωθεί σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου. Σε καμία περίπτωση. Εμείς λοιπόν στη βεβαιότητα του προπολογισμού προσθέτουμε και την αβεβαιότητα των νέων κανόνων και αφήνουμε ε, τους ε, γεωργούς μας μέσα σε ένα θολό τοπίο. Θα πρέπει να αποφύγουμε λοιπόν να βάλουμε τους ε, γεωργούς μας μέσα σε ένα τέτοιο άγνωστο τοπίο και ε, να τους γεμίσουμε βεβαιότητα για το μέλλον τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. κύριος Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να συγχαρώ καταρχάς τον συναδελφό μας, τον κύριο Χόφμαν, για το σχέδιο της έκθεσής του. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε καινούργια ΚΓΠ. Δεν χρειάζεται όμως να βιαζόμαστε, γιατί πρέπει αρκετά νωρί να ξέρουμε ποια θα είναι τα κονδύλια για να ξέρουμε τι θα κάνουμε το Γενάρη του 2021 να επιμείνω για την ανάγκη συνάφειας. Δηλαδή, να μην έχουμε μόνο τα κονδύλια για τους γεωργούς από αυτή την κοινή γεωργική πολιτική, γιατί έχουμε και το θέμα των διεθνών συμφωνιών. Και επιμένω, θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια στην στρατηγική όταν θα κάνουμε διαπραγματεύσεις με εταίρους παγκοσμίως δεν ωφελεί σε τίποτα να κάνουμε συμφωνίες για τα βοηθή τη στιγμή που οθούμε τους κτηνοτρόφους σε πτώχευση. Επίσης στο Omnibus θα πρέπει το δικαίωμα του ανταγωνισμού να συνοδεύεται από την ανάγκη οι γεωργοί να μπορούν να συμμαχούν, να συσπηρώνονται σε σχέση με τις βιομηχανικές μετατροπές που αφορούν και την ε, μεταποίηση. Επίσης υπάρχει μια ανάγκη. Εγώ στην εκλογική μου περιφέρεια δύσκολα μπορώ να εξηγήσω όλους τους βυζαντινισμούς της κοινή γεωργικής πολιτικής. Και για τον προϋπολογισμό ελπίζουμε να διατηρηθούν τα κονδύλια. Όμως για να διατηρηθούν τα κονδύλια δεν θα πρέπει μόνο να πείσουμε τους γεωργούς ότι δεν θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες, αλλά τους ίδιους τους Ευρωπαίους και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύμφωνο μεταξύ Ευρωπαίων πολιτών και Ευρωπαίων γεωργών που θα έχει στόχο τη διασφάλιση της ε, επάρκειας, της επισητιστικής αλλά και της διατήρησης, της διασφάλισης κοινών αγαθών ευρωπαϊκών για την υγεία, για το περιβάλλον, για το κλίμα και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι να κατανοήσουν τη διάρθρωση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Δηλαδή να έχουμε κονδύλια της κοινή γεωργικής πολιτικής που θα προορίζονται στην έρευνα. Αν θέλουμε να καταργήσουμε κάποιες βλαβερές ουσίες, τότε θα πρέπει ακριβώς να επενδύσουμε στην έρευνα ώστε να προτείνουμε στους γεωργούς υποκατάστατα όταν απαγορεύουμε κάποιες ε, βλαβερές ουσίες. Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα διασφαλίσεων το οποίο θα είναι ενθαρρυντικό και όπως προτείνει ο εισηγητής θα πρέπει να εγγράφεται στον κάθε ετήσιο προπολογισμό ώστε να υπάρχουν οι απαραίτητες για τους γεωργούς και τέλος να τονίσω την ανάγκη αποφυγής της επαναθνικοποίησης της κοινή γεωργικής πολιτικής γιατί έχουμε αυτά τα τρία κύρια στοιχεία κοινή, γεωργική, πολιτική και το τι σημαίνουν. Ευχαριστώ. Συγχωρέστε με, αλλά έδωσα περισσότερο χρόνο στον πρόεδρο της Επιτροπής Προπολογισμών. Ελπίζω να είστε κι εσείς ε, το ίδιο και νεόδρο σε θα μιλάω στη δική σας Επιτροπή. Κύριε Μπόκοβιτς, ε, ζητώ συγγνώμη και ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστούμε τον κύριο Ντόφμαν για αυτό το σχέδιο έκθεση. Συμφωνώ με όλες τις αρχές που οδηγούν στην απλούστευση και τη δική κατανομή. Αλλά εσεί αναφέρατε πώς μπορεί να γίνει όλο αυτό μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των γεωργών. Όλα κινούνται προ τη σωστή κατεύθυνση. Τα υποστηρίζω τώρα για το greening. Πιστεύω ότι μπορεί να επεκταθεί περισσότερο ε, στο περιβάλλον στη Γεωργία, διότι γνωρίζουμε ότι η πράσινη γεωργία είναι επίσης σημαντική και για το περιβάλλον. Τώρα, όσον αφορά για τη μεταβατική περίοδο, όσον αφορά τη μεταβατική περίοδο, θεωρώ ότι η περίοδος που δίνεται είναι υπερβολική. Θέλω να τονίσω ε, τρία πράγματα στις ε, παραγράφους 15, 16 και 19, χωρίς τους νέους γεωργούς χωρίς τα δικά τους εισοδήματα θα πάψουν να υπάρχουν στην ε, Ήπεθρο αποκλείεται να γίνει ψηφιοποίηση ε, στην Γεωργία και χωρίς ε, την ψηφιοποίηση η Γεωργία θα βρεθεί σε δινή θέση και όλη η ανάπτυξη της υπαίθρου στο σύνολό της επίσης όλα αυτά ε, αφορούν ε, θέματα ενεργειακά, τεχνολογικά. Δεν χρειαζόμαστε μόνο έξυπνες πόλεις, αλλά και έξυπνα χωριά, έξυπνη εξοχή, έξυπνη ύπεθρο. Ε, όσοι από εσά θα συμμετέχετε στην Επιτροπή για τα λοιπάσματα, μπορείτε να πάρετε το λόγο τώρα ο κύριος Ταραμπέλα και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαιρετίζω την δουλειά του συναδέλφου, παρόλο που θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε το θάρρος να πάμε πέραν της προοπτικής του 2027 δηλαδή πι δελτα και να πάμε σε ένα μακρόπνο σχέδιο που θα αφορά επενδύσεις τους νέους γεωργούς σε βάθος δεκαετιών. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερη σταθερότητα, θα πρέπει να έχουμε πιο δίκαιη κατανομή της ε, δημόσια στήριξη. Επίση, θα πρέπει να έχουμε περισσότερη βιωσιμότητα ακριβώ για να διασφαλίσουμε το μέλλον των νέων γεωργών, ανδρών και γυναικών. Και θα πρέπει επίση να ασχοληθούμε με την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η Επιτροπή των Περιφερειών που θέλω να διαφημίσω εδώ και η οποία δεν αναφέρεται και τόσο συχνά είχε μια έκθεση του συνάδελφου Γκρό, σοσιαλιστή, ο οποίο, ναι, εντάξει, το καταλαβαίνω, θα έχετε αντιρρήσει, αλλά έκανε πολύ καλή δουλειά εκ μέρου των σοσιαλιστών για αυτό το θέμα και μίλησε, α πούμε, για τι ελλείψει, μίλησε για τι ποσοστώσει στα γαλακτοκομικά και τόνισε το ότι οι, οι κτηνοτρόφοι όταν έχουν χαμελές ε, τιμές στα προϊόντα τους, θα πρέπει να αναζητήσουν νέες αγορές. Οπότε πάνε αλλού. Και ποιος ωφελείται, οι πολυεθνικές. Και κάτι άλλο. Θα πρέπει να περάσουμε από τη στασμεύση στις συμφωνίες, στις συμβάσεις. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις δηλαδή οι οποίες θα πρέπει να είναι εφαρμόσιμες και αποδεκτές από τον κόσμο της Πέθρου, από τους γύρους και πρόεδρε, να καταλήξω λέγοντας ότι θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τότε όριο βεβαίω στις ενισχύσεις, όχι όμως σε σχέση με την παραγωγή, αλλά σε σχέση ας πούμε με την ε, εργασία ανακτάριο. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που κάνουν και άλλοι μεγάλοι διεθνεί ε, ε, παράγοντες που ακολουθούν άλλα κριτήρια, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομη επειδή ο συνάδελφος ο Αρτουή είπε πολλά από αυτά που ήθελα να πω και εγώ. Να σας πω ότι συμφωνούμε σε αρκετά σημεία και ευχαριστούμε τον κύριο Ντόρφμα για τη δουλειά που έκανε. Να αφιστήσω μόνο την προσοχή σας στο γεγονό ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα ψηφίσει μια έκθεση τέλη του Απρίλη που θα παράσχει κάποιες κατευθυντές γραμμές όσον αφορά τα θέματα του περιβάλλοντος που αφορούν την επόμενη ΚΓΠ. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει μια συνάφεια στην δουλειά που κάνουμε εδώ και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, ώστε πραγματικά η κοινή γεωργική πολιτική να εξυπηρετήσει, να υπηρετήσει τους πολίτες και τους γεωργούς. Γεωργούς που έχουν απομιστεί ε, με το έργο της ε, διατροφής όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ θα ήθελα να τονίσω και εγώ το θέμα του περιβάλλοντος. Το... Είχαμε μία πρόσφατη μάλλον έκθεση που αφορούσε το πρασίνισμα της κοινής πολιτικής που όμως δεν παρουσιάζει απτά αποτελέσματα και πλεονεκτήματα για το περιβάλλον. Είναι λοιπόν κρίμα που αυτή η κατά τα άλλα εξισορροπημένη έκθεση δεν είναι ε, αρκετά ισχυρή σε κάποια ζητήματα. Εντάξει, αναφέρουμε το τι θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι Γεώργοι όσον αφορά τι μεταβολέ των τιμών κτλ. Αλλά αυτά τα απτά προβλήματα εδώ και χρόνια έχουν αφήσει τη θέση του σε άλλα προβλήματα, πολύ πιο σοβαρά. Το κόστος, ας πούμε, παραγωγής, ε, το θέμα των εκμεταλλεύσεων και των μεγάλων επιχειρήσεων. Όλα αυτά αποσιωπούνται στην έκθεση. Οι άμεσες ενισχύσεις και πληρωμές. Τι γίνεται με όλα αυτά, τα οποία είναι απαραίτητα για την επιβίωση των κάποιων εκμεταλλεύσεων. Επίσης δεν αναφέρεται ότι τα δεδομένα που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παροχημένα γιατί δεν λαμβάνει υπόψη τους κάποιες πρόσφατες κρίσεις. Και τέλος, οι συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών δεν χαράζονται με ξεκάθαρο τρόπο όπως η ΣΕΤΑ και η Μερκοσούρ και ο μηχανισμός προστασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη του συμφωνίες όπως αυτές που είχαμε τη Γεωργία, την Ουκρανία, το Μαρόκο κτλ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εμεί που θέλουμε να κρατήσουμε ή να ενισχύσουμε τον προπολογισμό της ε, ΚΑΠ πρέπει να είμαστε και έτοιμοι να διορθώσουμε τα λάθη της και τις ανεπάρκειες. Έτσι λοιπόν σε εκθέσεις όπως αυτή που γίνεται λόγος για ανοχή καταστάσεων στην Ιρλανδία παραδείγματι είναι 17.000 ευρώ το χρόνο ο μέσος όρος ενώ μια μικρή εκμετάλλευση μπορεί να παίρνει ε, πολύ λιγότερα ποσά. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να εξασφαλίσουμε. Τι έγινε τώρα, δεν με καταλαβαίνετε. Πρέπει λοιπόν να πείσουμε και έχουμε και άλλα ζητήματα σοβαρά να λύσουμε. Κλιματική αλλαγή. Ενώ ταυτόχρονα λέμε ότι θέλουμε να υποστηρίξουμε εμπορικέ συμφωνίε οι οποίε φέρνουν προϊόντα από την άλλη άκρη του πλανήτη ε, ενώ έχουμε πολύ καλύτερη ποιότητα προϊόντα παραγόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν δεν λύνει το πρόβλημα, μάλλον το επιδεινώνει. Καπ, λοιπόν, χωλαίνει. Δεν μπορούμε να τη σώσουμε εάν δεν δώσουμε μια σοβαρή απάντηση στα προβλήματά της και δεν πείσουμε και τον πολίτη για την διατήρηση και ενίσχυση, για την ανάγκη διατήρηση και ενίσχυση των επιπέδων του προπολογισμού και αυτό με επίλυση, με αντιμετώπιση των ανισοτήτων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον συγχαρώ τον κύριο Ντόρφμαν για την έκθεσή του. Μια γενική παρατήρηση για τις αντιδράσεις και τους τομείς που καλύπτει η Επιτροπή μας. Συνήθως ε, έχουμε να κάνουμε με μια αντίδραση η οποία μπορεί να εκφράζει και το φόβο ότι θα αλλάξει ριζικά η ΚΑΠ. Γιατί λοιπόν να μην ε, κάνουμε ένα βήμα προς τα πίσω, να πάρουμε απόσταση δηλαδή και να αναλογιστούμε πρώτα απ' όλα τι θέλουμε από μια κοινή γεωργική πολιτική. Έχει επταετή διάρκεια. Καταρχάς μην το ξεχνάμε, θα χρειαστούν κάποια χρόνια για να ε, ληφθούν αποφάσεις Άρα μιλούμε για την έναρξη εφαρμογής σε καμιά δεκαετία σε έναν κόσμο που αλλάζει. Τι στόχους έχουμε λοιπόν, τι θέλουμε να επιτύχουμε με την Κούγουπο. Ας μην μιλάμε για πυλώνες, ας μην μιλάμε για ε, ενίσχυση, ας μην μιλούμε για ε, διακύμανση. Ας δούμε τι στόχους θέλουμε να υπηρετήσουμε. Δύο είναι οι σαφείς στόχοι. Πρώτον, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του γεωργού, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε γεωργούς, οι οποίοι την ενίσχυση στο εισόδημα την ε, χρησιμοποιούν μόνο και μόνο για την επιβίωσή τους. Δεν ε, επενδύουν στις εκμεταλλεύσεις τους για να τους εξασφαλίσουν ένα μέλλον. Ε, άρα λοιπόν θα πρέπει να λύσουμε όποια προβλήματα μπορεί να εμφανιστούν με μια κρίση, με ένα ταμείο κρίσεων, το οποίο πάλι ενισχύει την εξάρτηση του Γεωργού. Πρέπει να βρούμε λύσεις λοιπόν, λύσεις ευφυής, με εργαλεία, με καλύτερη οργάνωση, με διαχείριση κρίσεων, έτσι ώστε να είμαστε λιγότερο εξαρτημένοι από τα χρήματα που δίνουν οι Βρυξέλλες. Και το άλλο θέμα, το ότι πρέπει ο γεωργικός τομέας να λειτουργεί ικανοποιητικά, ώστε να προσφέρει τα προϊόντα όπως τα θέλουμε. Μερικές φορές πρέπει η ελεύθερη αγορά να καλύπτει τις ανάγκες και μερικές φορές ε, όχι. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν, πρόεδρε ευχαριστώ τον κύριο Ντόρφμαν. Και μια και μιλάμε μερικέ μέρε μετά από την ημέρα τη της γυναίκα, τη μητέρα μάλλον στην Αγγλία, θα ήθελα να ευχαριστώ τη μανούλα μου που με έφερε στον κόσμο. Νομίζω λοιπόν ότι Πρέπει να συστήσουμε ποιο θέλει να μπει στο γεωργικό χώρο, να εργαστεί ω αγρότη και να μείνει αγρότη. Για να το καταφέρουμε αυτό, να μείνουν αγρότε, είναι απαραίτητο να του προσφέρουμε και έντιμη ανταμοιβή και αποζημίωση του κόπη του, αλλά και την αναγνώριση την ψυχολογική υποστήριξη για μια ε, και κατανομή επίσης θα μιλήσω που απαιτείται που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή και πάντως όχι στην Ιρλανδία ένα ισότιμο σύστημα καταβολής αμοιβών για το δημόσιο αγαθό της βιοπικιλότητας, του περιορισμού της κλιματικής ε, αλλαγής που εξασφαλίζει ο Γεωργός. Και αυτό θα μας φέρει σε επίπεδο κάλυψης των εισοδηματικών αλλαγών των Γεωργών. Δεν νομίζω βέβαια στο θέμα των γενεών, για να αναφερθώ, ότι έχουμε ποτέ εκφράσει τόσο προσβλητικά λόγια σε κάποιον εκπρόσωπο άλλου επαγγελματικού κλάδου πέραν αυτού των γεωργών, ρωτώντας τον γιατί δεν θες να πας να, να ξεκινήσεις μια δουλειά που στο τέλος ε, του μήνα θα σου αφήνει λιγότερα χρήματα από όσα έχεις επενδύσει, γιατί αυτό κάνουμε τους γεωργούς, αλλά κομμωτές ή άλλους δεν ρωτάμε αν θέλουν να, κάνουν, να, να ξοδέψουν έτσι τα χρήματά τους. Τώρα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτού που πρέπει να φύγουν στη σύνταξη, πρέπει να καλύψουμε αυτού που θέλουν να μπουν στην γεωργική δραστηριότητα, αλλά πρέπει και να εξασφαλίσουμε χώρο για του νέου αυτού ε, γεωργού. Και πολλά είναι τα καλά της έκθεσης. Ε, η αναθεώρηση των ιστορικών πληρωμών είναι μια πολύ καλή ιδέα. Είναι πολύ καλή ιδέα τη στοχευμένη τη υποστήριξη στι μικρέ οικογενειακέ εκμεταλλεύσει. Σε ένα σημείο όμω με προβληματίζει η έκθεση εκεί που αναφέρεται στην ανάδειξη νέων προκλήσεων στο παγκόσμιο εμπόριο. Μα δεν είναι η ανάδειξη. Εμεί το πρόβλημα το δημιουργούμε οι ίδιοι. Με αυτέ τι εμπορικέ συμφωνίε προξενούμε το πρόβλημα. Επομένω, εάν αναδύονται προβλήματα, σταματήστε τα μην τους επιτρέπεται να αναδύονται, ώστε να μην εξαντλούνται και οι γεωργοί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. το ζήτημα της εκμετάλλευση των γεωργικών προϊόντων στο πλαίσιο της ΚΑΠΑ και η επαρκής αμοιβή των γεωργών, η συνοχή, η εδαφική. Όλα αυτά είναι σημαντικά θα πρέπει να προχωρήσουμε σταδιακά στη, προς ένα σύστημα άμεσων ενισχύσεων προς τα κράτη-μέλη. Οι Ευρωπαίοι Γεωργοί δεν καταλαβαίνουν τη διαφορά της στήριξης ε, του πυλώνα 1 μεταξύ πιο πλούσιων και λιγότερο πλούσιων χωρών. Τα κριτήρια ε, ιστορικής αναφοράς ε, θα πρέπει να τα ζητήσουμε προσεκτικά. Θα πρέπει να προβλέψουμε μία μετάβαση. Πρέπει να προωθήσουμε την αλλαγή που θα γίνει ε, στους γεωργούς και θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες προθεσμίες διότι δημιουργείται αβεβαιότητα ε, μεταξύ των γεωργών και θα πρέπει να ε, δημιουργήσουμε και ένα αποθεματικό κρίση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώνα, ειδικότερα για τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης θα πρέπει να δίνουμε ευελιξία στα κράτη-μέλη όσον αφορά την κινητοποίηση. Είναι πολύ σημαντικά ε, η εισαγωγή προϊόντων από τρίτες χώρες ε, ε, αλλά πρέπει να τηρούν τις ίδιες, τα ίδια πρότυπα. Θα πρέπει όλες οι ευρωπαϊκές περιοχές να λαμβάνονται υπόψη, ακόμη και αν απομακρυσμένες. Θα πρέπει να βασιστούμε στα άριστα ε, αποτελέσματα που είχαμε στο πλαίσιο της Επιτροπής ε, Γεωργίας ε, είχαμε κάποιο κονδύλο για το ΠΟΖΕΙ και θέλουμε να ληφθούν όλες οι ιδέες μας υπόψη και ελπίζουμε την Τετάρτη να ληφθούν υπόψη. Η ΚΑΠ δεν χρειάζεται τεράστιε τροποποίησεις Έχουμε εξαλλού λίγο χρόνο. Χρειάζεται σταθερότητα, προβολή, fair play, απλούστευση, επισητιστική ασφάλεια και μείωση του διοικητικού φόρτου. Ευχαριστώ. Euh, ναι, δεν θα ε, ξεκινήσω ξανά τις μεγάλες συζητήσεις ε, για την επιστημιστική κυριαρχία, το ζήτημα του κλίματος ε, και τις ελεύθερες συναλλαγές που είναι πρόβλημα. Θα μιλήσω για πράγματα που δεν έχουν υποθεί ακόμα. Πρώτον, όσον αφορά το ζήτημα μεταξύ προπολογισμού και γεωργικής πολιτικής, ο μεγάλος κίνδυνος σήμερα που διαβλέπω εγώ είναι ότι έχουμε πάρα πολύ όμορφες προτάσεις με τις οποίες συμφωνώ γιατί τις έχουμε προτείνει εδώ και καιρό, ε, το ανώτατο όριο το, στις ενισχύσεις, το capping. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ σήμερα είναι ότι όταν η Επιτροπή μας μιλάει για επιβολή ανώτατων όριων στις ενισχύσεις, πίσω από αυτό ο στόχος υπάρχει η μείωση του μεγέθους των ενισχύσεων, του μεγέθους της ΚΑΠ. Οπότε η πρόταση αυτή αποσκοπεί όχι στο καλύτερη κατανομή για να χρηματοδοτηθούν και άλλες πολιτικές, αλλά στη μείωση της ΚΑΠΟ. Οπότε αυτό είναι το θέμα τη συζήτηση. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο, όταν μιλάμε για κατανομή μεταξύ κρατών μελών, των άμεσων ενισχύσεων για του γεωργού στο πλαίσιο του πρώτου πυλώνα, τότε αντιληφθήκαμε ότι αν περιμέναμε του κανόνες έτσι όπως έχουν σήμερα θα έπρεπε να 30 χρόνια για να εξισωθούν οι ενισχύσεις μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης στο στόχο πρέπει να έχουμε εναρμόνιση τουλάχιστον το, το πολύ εντό δεκαετία μεταξύ Δύση και Ανατολή τη Ευρώπη. Αλλιώ θα δημιουργήσουμε μια κρίση εντό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία. Παρεμπιπτόντω τώρα προκύπτει το ζήτημα του πώ θα προτείνουμε βοηθήσει, ε, βοήθεια και αποθεματικό κρίση όταν γνωρίζουμε ότι η διάλυση των εργαλείων παραγωγής και σκέφτομαι το αγαλακτοκομικά τώρα θα διοδηγήσουν σε μια κρίση που ήδη είναι ορατή μέσα στον επόμενο μήνα, στο επόμενο δίμηνο. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση επικίνδυνη και θα πρέπει να συζητήσουμε σε βάθος, αλλά δεν μπορούμε να συζητάμε χωρίς σε επίπεδο προϋπολογισμού να έχουμε μια οικονομική επένδυση, ε, συγγνώμη, βεβαίωση, εγγύηση διατήρηση του επίπεδου ενίσχυση, όχι μόνο στο, εδώ στο κοινοβούλιο που συζητάμε, σε επίπεδο κρατών μελών. Ναι. Και εγώ να ευχαριστήσω τον κύριο Ντόρμαν τον εισηγητή γιατί έχει κάνει μια εργασία την οποία σε γενικές συμμερίζομαι. Να πω και κάποια πράγματα που δεν αναφέρθηκα μέχρι τώρα. Στον ελάχιστο χρόνο που έχουμε θα πρέπει να θέσουμε στην Κομισιόν κάποια ζητήματα και θα πρέπει να υποφεληθούμε της ευκαιρίας για να στηρίξουμε την καινοτομία, την τεχνολογία, την ανάπτυξη που σημειώνεται στη Γεωργία. Νομίζω θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερα προσοχή στην ολοκληρωμένη Γεωργία. Κάτι με το οποίο ασχολούνται οι Γεωργοί και εμεί ακόμα δεν έχουμε αναγνωρίσει αυτές τις προσπαθίες τους. Νομίζω λοιπόν θα μπορούσαμε να προσανατολίσουμε τη δουλειά μας που θα κάνουμε άμεσα στο μέλλον προς τα εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πρόταση έκθεσης και νομίζω ότι στην έκθεση μας θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν ενισχύσει πανευρωπαϊκέ, ευρωπαϊκού χαρακτήρα που θα επιτρέπουν στι χώρε μέλη να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένε καταστάσει. Θα πρέπει λοιπόν οι χώρε μέλη να συνεχίσουν να διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα χωρί να προηγηθούν διαπραγματεύσει. Η κοινή πολιτική θα πρέπει για την νέα περίοδο να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει και εξωτερικούς παράγοντες. Νομίζω ότι οι πληρωμές στον πρώτο πυλώνα είναι διαφορετικές από τις πληρωμές στον δεύτερο. Γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να ακολουθήσουμε και διαφορετική προσέγγιση. Κυρίως εδώ έχουμε να κάνουμε με την εξωτερική σύγκληση. Μετά για τις αγορές θα πρέπει να υπάρχει η απαραίτητη προσφορά σε, περιόδου σε περίοδους κρίσης ώστε να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι θα πρέπει να υπάρχουν και τα κατάλληλα χρηματοοικονομικά εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ακραίες κρίσεις που έχουμε καμιά φορά. Και τέλος, θα ήθελα να περιληφθούν προγράμματα που θα αφορούν την μελισουργία και τις μικρομεσαίες επιχείρησεις που εργάζονται στον τομέα αυτό. Εγώ θα εργαστώ ε, πολύ σε αυτά τα θέματα και ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση του. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, να πω και εγώ ότι ευχαριστούμε τον εισηγητή για την έκθεσή του, αλλά κύριε Ντόφμαν, ανησυχώ πολύ για το άρθρο 13 για τις ε, ενισχύσεις οι οποίες αναφέρεται ότι θα λαμβάνουν υπόψη του κόστη παραγωγής, ε, κοινωνικονομικές συνθήκες που επικρατούν στι χώρες μέλη κτλ. Εγώ συνάδελφοι κατάγομαι από την Ανατολική Ευρώπη και εμείς υποφέρουμε επειδή έχουμε πολύ χαμηλότερες πληρωμές σε σχέση με άλλες ε, χώρες της Ένωσης τη στιγμή που είμαστε υποτίθεται ισότιμοι εταίροι. Πρέπει να ληφθούν υπόψη Βεβαίω οι διαφορέ μεταξύ χωρών μελών, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι πέραν του 2020 θα συνεχίσουμε να έχουμε πολύ σημαντικέ, πολύ υψηλέ υψηλές διαφορές στις πληρωμές μεταξύ Ανατολική και Δυτική Ευρώπη. Θεωρώ λοιπόν ότι έστω και αν δεν συμφωνούν όλοι, θα πρέπει να, συνοδεύεται, να συνοδεύονται αυτές οι ενισχύσεις με την παραγωγικότητα στη Γεωργία. Γιατί όλα αυτά που ακούγονται ότι εμεί δαπανάμε πάρα πολλά χρήματα στην Γεωργία και για το κάνουμε αυτό, φαίνεται ότι τελικά δεν ισχύουν. Και θα ήθελα να καταλήξω λέγοντα το εξή. Βλέπω ότι κάποιε χώρε ρωτάνε το... και λένε γιατί χρειαζόμαστε τόσα πολλά χρήματα. Αν κάποιο λοιπόν καταναλώνει συγκεκριμένα αγαθά σήμερα τα ένα κόστο που θα μπορούσε να ήταν πολύ ψηλότερο διαφορετικά αν δεν είχαμε αυτέ τι ενισχύσει. και θα μπορούσαμε να είχαμε σε χειρότερη, στη χειρότερη περίπτωση και εισαγωγέ σε πολύ επικίνδυνε από άλλε χώρε. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα για μένα είναι αν μπορούμε να έχουμε μια απλή εφαρμογή των προτάσεων. Ξεχνάμε ότι στο επίκεντρο των ενδιαφέροντό μας είναι ο Γεωργός ε, σταδιακή μείωση και ανώτερα επίπεδα θεωρώ ότι θα πρέπει να αφαιθούν στα κράτη-μέλη. Ένα παράδειγμα, 30 εκτάρια ε, έκτασης εκμεταλλεύσης στην ε, Βαβαρία μπορεί να θεωρούνται σε άλλες περιοχές μεγάλα, σε άλλες χώρες δηλαδή μεγάλη έκταση, σε άλλες μικρές. Εν πάση περιπτώσει πρέπει να βρούμε μια καλή λύση και πρέπει νομίζω αυτή η λύση να δοθεί από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Δεν μπορεί να τα ρυθμίζει η Ευρώπη. Ο κύριος Στόρφμαν επίσης μιλάει για μεταβατικές διατάξεις μέχρι ότου ετοιμαστεί και η υλοποίηση της ε, μεταρρύθμισης βεβαίως μπορεί απλώς να παρατεθεί το όμνιμπους, ο κανονισμός όμνιμπους. Νομίζω ότι μπορεί αυτό να προσφέρει την ασφάλεια που χρειάζονται οι γεωργοί ω μετάβαση. Σας ευχαριστώ. Κυρία Κατάινεν. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον κύριο Ντόρφμαν. Είναι πολύ καλή και ισορροπημένη πρόταση. Εδώ έχουμε να κάνουμε με το εισόδημα των γεωργών. Αυτό πρέπει να λάβουμε πάνω από όλα υπόψη και νομίζω το καταφέρνει η πρόταση του κυρίου Ντόρφμαν. Κάποιες ε, βελτιώσεις θα πρότεινα για τον ε, δεύτερο πυλώνα που αναφέρει ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εθνικά δεδομένα. Οι άμεσες ενισχύσεις όμως βρίσκονται αντιμέτωπε με διαφορές μεταξύ εθνικών ε, διαφορών. Επίσης θα πρέπει να κοιτάξουμε όταν μιλούμε για μικρές ε, εκμεταλλεύσεις, να μην πέσουμε στην παγίδα, να καλύπτουμε και να ψωτεύουμε ιονή παραγωγούς ή παραγωγούς. Πρέπει να κοιτάξουμε ποιες είναι πραγματικά οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και βέβαια και τους νέους γεωργούς να στηρίξουμε. Επίσης θα ήθελα ως νέο, νέο μέλος της Επιτροπής να προσκαλέσω τον κύριο Ντόρφμαν και μια αντιπροσωπεία της Επιτροπής ε, Γεωργίας στην πατρίδα μου τη Φιλανδία για να συζητήσουμε με ε, τα, θέματα αυτά όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Κύριος Νεύκοφ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για να μπω στην ουσία της συζήτησης. Ε, σημαντικό θέμα είναι η αρπαγή γεών. Για ορισμένες χώρες τουλάχιστον ένα τεράστιο πρόβλημα που εμποδίζει την, ανάδειξη, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από νέου γεωργούς. Πρέπει σε αυτό να δοθεί μία λύση, μία λύση ισορροπημένη μεταξύ της προσφοράς ενισχύσεων αλλά και της διαφύλαξης της δραστηριότητας. Ίσως πρέπει πάνω απ' όλα να ελέγξουμε αν είναι γνήσιος παραγωγός αυτός τον οποίο ενισχύουμε ή να προσφέρουμε την ενίσχυση ως ανταμοιβή για την ε, διατήρηση δημιουργία ανένθεσεων εργασίας. Αγορές, ε, κοινέ αγορές προϊόντων, οργανωσης αγορών. Ε, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είναι κοινά τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο γεωργός, η κλιματική αλλαγή, οι επιζωοτίες, άλλες νόσοι. Και έτσι θα έλεγα ότι ανάμεσα στην ε, Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη ε, Φινλανδία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα δεν μπορώ να δικαιολογήσω γιατί υπάρχουν τόσες διαφορές στις ενισχύσεις. Πρέπει να είναι ίδιες οι ενισχύσεις. Και αυτό περιμένουν και οι Ευρωπαίοι σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι θα πρέπει να ανταμείβουμε τους αγρότες και όχι να τους εμποδίζουμε. Σας, συμφωνώ με εσά ω ε, Πρόεδρο τη ε, Επιτροπή Προπολογισμών. Οι Γεωργοί παίζουν σημαντικό ρόλο και σε άλλε οικονομικέ δραστηριότητε και σε άλλου τομεί. Κοιτάξτε την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα, για τα πτηνά, για τα οικοσυστήματα. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά. Συμμετέχουν και οι γεωργοί. Πρέπει να αναγνώσουμε τον οριζόντιο χαρακτήρα του και πώ ε, επηρεάζουν όλου του τομεί. Ναι, συμφωνώ, χρειαζόμαστε περισσότερα προϊόντα, περισσότερα περισσότερο τρόφιμα, αλλά και οι γεωργοί πρέπει να αμείβονται επαρκώ. Πρέπει λοιπόν να τα συμφιλιώσουμε αυτά. Μιλάμε τώρα για κοινή αγροτική πολιτική. Εγώ είμαι υπέρ των οικογενειακών γεωργικών επιχειρήσεων. Οι πολυεθνικέ ούτω ή άλλω θα ζήσουν. Αυτέ αγοράζουν τι γέε ω ε, επενδύσει. Θα, εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε τη, να υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξη της υπαίθρου και ότι οι γεωργοί θα συνεχίσουν να υπάρχουν. όλα αυτά μπορούν να συνδεθούν και με άλλου τομεί και να χρησιμοποιήσουμε εκεί τι επενδύσει ε, που λέει ο Γιούνκερ. Ε, στον πυλώνα 1, στον πυλώνα 2 λέμε και αναρωτιούνται στον χώρο μου τι θα γίνει με όλα αυτά. Πρέπει να αρχίσουμε να ανταμείβουμε του ε, γεωργού για τι προσπαθίε του και όχι να του βάζουμε τρικλοποδιέ. Και φυσικά θα πρέπει να δούμε και την ευρύτερη εικόνα. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στα σταυροδρόμοι. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εδώ έχει γίνει καταπληκτική δουλειά, το βλέπω. Πρέπει απλώς να επεξεργαστούμε λίγο περισσότερο το κείμενο για να το βελτιώσουμε. Εγώ έχω φέσει τακτικά με γεωργούς, συζητούμε τα διάφορα προβλήματά τους. Από τη μια λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση για την επανεθνικοποίηση. Αλλά ιδιαίτερη ανησυχία, ιδιαίτερη ανησυχία προξενεί το γεγονός ότι δεν εγγυάται αυτή ότι θα κλείσει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών γεωργών. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν. Πρέπει η αγορά να εξασφαλίζει, στην αγορά να εξασφαλίζουμε ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού. Κάτι ακόμη. Το οποίο δεν είναι και αιτιολογημένο πιστεύω. Δεν είναι καλό, δεν είναι σωστό να χρειάζεται να πηγαίνουν να δουλεύουν ως εργατικά χέρια στη συγκομιδή ε, εργάτες από τα ανατολικά κράτη αλλά να μην μπορούν να επιβιώσουν στις ίδιες τους χώρες. Γι' αυτό λοιπόν αυτό το χάσμα πρέπει να καλυφθεί. Και αντίστοιχα και στο σημείο 13 θα ήθελα να υπάρξει διόρθωση του κειμένου. Να υπάρχουν οι ίδιες συνθήκες, ε, αλλά πρέπει να πούμε και πώς θα εξασφαλιστούν αυτές. Πρέπει να πούμε με ξεκάθαρο τρόπο ότι πρέπει να έχουμε ισότιμες συνθήκες. Πώς θα οριστεί δηλαδή η τιμή σε ένα κατάστημα. Ε, μπορεί κάποιος να πάει και να πει είναι πολύ ακριβή η τιμή, αλλά να έχει ο άλλος φτυσίαιμα για να το παράγει το προϊόν. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και εγώ εκτιμώ την προσπάθεια του αδελφού Ντόρφμαν αλλά συμφωνώ με τους αδελφούς για τι ενισχύσει. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ των χωρών μελών ώστε να εξαλείψουμε τι οικονομικέ και κοινωνικέ ε, διαφορέ που υπάρχουν. Νομίζω ότι οι ενισχύσει θα πρέπει να κατανείμονται με τρόπο δίκαιο και ισότιμο μεταξύ των χωρών μελών. Επίσης πιστεύω ότι θα πρέπει να μιλήσουμε για το γεγονό ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πολύ σοβαρή πρόκληση, τη γύρανση του πληθυσμού της δηλαδή. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να στηρίξουμε τους νέους γεωργούς για το μέλλον. Και Νομίζω θα πρέπει να αποτελεί μια προτεραιότητά μας αυτό. Έχουμε ακούσει διάφορα προς την κατεύθυνση αυτή, αλλά δεν έχουμε γενεακή αλληλουχία στη Γεωργία και αυτό θα αποτελέσει ένα σοβαρό πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους νέους ώστε να πάνε να ζήσουν στην Ήπεθρο και ενδεχομένως να ασχοληθούμε τη Γεωργία, να αρχίσουν να δημιουργούν γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίες βέβαια θα πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες τεχνολογίες και στις νέες συνθήκες και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικότητα αυτών των νέων ανθρώπων και σε άλλες μορφές που αφορούν τη γεωργία όπως οικοτουρισμό, γεωργικό τουρισμό, ανάπτυξη της υποδομής και παροχή άλλων υπηρεσιών επίσης, ώστε να πιστούν οι νέοι να πάνε να ζήσουν στις υπαίθρους και να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη γεωργία. Ευχαριστώ. Κύριε Μακίνες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Με ενδιαφέρον άκουσα τις διάφορες απόψεις. Έστειλα σε 7 διαφορετικές οργανώσεις την πρόταση έκθεσης και δεν υπήρχε συνένεση μεταξύ τους για την, τον περιχώμα της έκθεσης. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να καταθέσουμε πάρα πολλές τροπολογίες στην πρόταση αυτή, να δαπανίσουμε χρόνο, ενέργεια και δύναμη, να συζητήσουμε με το Συμβούλιο και τελικά να χάσουμε σε πολλά σημεία. Θα ζητήσω λοιπόν να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να σκεφτούμε και να δούμε ακριβώς τι εννοούμε με το οικογενικές εκμεταλλεύσεις, γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Υπάρχουν διάφορες μορφές αυτών των εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη. Ποικίλει το μέγεθος, ποικίλουν τα χαρακτηριστικά τους μεταξύ των χωρομελών. Πρέπει να το δούμε. Μετά, για τα ανώτατα όρια, για το κάπινγκ. Πρέπει να το δούμε αλλά δεν θα πρέπει να το αποφασίσουν αυτό οι χώρε μέλη. Πρέπει να είναι αντικείμενο απόφαση σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Και για τους νέους γεωργού. νομίζω ότι έχουμε κάνει καλή δουλειά, πρέπει όμως να κάνουμε περισσότερα και να κάνουμε κι άλλα για να τους βοηθήσουμε μέσω διαφορών παρεμβάσεων. Επίσης, θα ήθελα να δω και τις προτάσει της Κομισιόν για την διατροφική αλυσίδα ένα πολύ σημαντικό ζήτημα αυτό για τους Γιώργου. Εξού σημαντικό με την κοινή πολιτική. Ανησυχώ όμω, επειδή όπω λέγαμε προηγουμένω, θα καταθέσουμε πολλέ τροπολογίε για την έκθεση και δεν θα στείλουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς την Κομισιόν η οποία μπορεί να αποφασίσει κάλλιστα να αγνοήσει τι δικέ μα θέσει για αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι η νομοθετική πρόταση για την διατροφική αλυσίδα θα είναι έτοιμη το αργότερο τον Απρίλιο. Κομισιόν, κύριε Ναγιέλ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Έχει περάσει και η ώρα. Είναι αργά. Καλωσορίζουμε την έκθεση αυτή του κύριου Ντόρφμαν πολύ σημαντική η αξία της για τις μελλοντικές μας ομοθετικές προτάσεις και από ό,τι βλέπω όπως αναφέρει και η ανακοίνωσή μας του Νοέμβρη επηρεάζει πολύ τις προθέσεις μας. Πρέπει να συζητήσουμε και το νέο τρόπο επίτευξης όλων αυτών των κατευθυντήριων γραμμών που θα αφορά ενδεχομένω ίσως όχι όλους τους ε, πυλώνες της κοινή γεωργικής πολιτικής. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με την ε, ανάπτυξη της υπαίθρου και με άλλα ζητήματα. Κατέγραψα κυρίω, κυρίως δύο ζητήματα ανησυχίας. Η επανεθνικοποίηση της κοινή γεωρικής ε, πολιτικής και η να σας διαβεβαιώσω ότι δεν έχουμε πρόθεση να επαναεθνικοποιήσουμε την κοινή πολιτική. Αυτό που έχουμε κατά νου είναι να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις ώστε αυτή η πολιτική να είναι πραγματικά κοινή. Νομίζω ότι για πρώτη φορά βλέπουμε ότι υπάρχουν κοινά, κοινοί στόχη για το, και κοινή προσέγγιση για το πώ θα μπορούσαν να επιτευχθούν αυτοί οι κοινοί στόχοι πανευρωπαϊκά. Και αυτό νομίζω ήδη είναι αρκετά ισχυρό συνδετικό στοιχείο τη κοινή γεωργική πολιτική, Αλλά βεβαίω υπάρχουν και άλλοι παράγοντε που αφορούν τι νομοθετικέ μα προτάσει και θα πρέπει βεβαίω να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μια αρκετά ισχυρή κυβερνητική δομή η οποία βεβαίω θα τα εφαρμόσει σωστά όλα αυτά σε όλε τι χώρε τη Ένωση. Και συνολικά νομίζω ότι έχουμε ένα πολύ καλό πακέτο στα χέρια μας ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, ενδεχόμενες κριτικές και για να διασφαλίσουμε το κοινό χαρακτήρα. Άκουσα επίσης ότι υπάρχουν ανησυχίες για αυτό το πρότυπο επίτευξης, το οποίο ενδεχομένω προκαλεί αμφιβολίες σε κάποιες χωρισμένες σε σχέση με τις ενισχύσεις στον πρώτο πυλώνα και τις ε, ε, επεμβάσεις σε περιφερειακό επίπεδο. Νομίζω ότι εμείς θέλουμε να υπάρχει προσέγγιση ε, του πρώτου πυλώνα για το εθνικό σε εθνικό επίπεδο και αντίστοιχα στο περιφερειακό. Νομίζουμε ότι αυτό γίνεται κάλλιστα και θεωρούμε ότι θα μπορούσε να γίνει ακριβώς και με αυτά προβλέπουμε όσον αφορά την κατανομή των εξουσιών και των αρμοδιοτήτων στις χώρες μέλη. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία ουσίας που θα ήθελα να αναφέρω. Βλέπουμε, ας πούμε, στο σχέδιο έκθεσης να αναφέρεται το θέμα των γενεών και των νέων γεωργών. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί επίσης ε, έμφαση στην διαχείριση του κινδύνου και επίσης άλλο ένα σημείο που μας αφορά αυτή τη στιγμή έχουμε τα εργαλεία ως πίμα του Omnibus για την διαχείριση του κινδύνου στο δεύτερο πυλώνα αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εργαλεία διαχείριση του κινδύνου θα πρέπει πραγματικά να αφορούν και τον πρώτο πυλώνα τη ε, κοινή ε, αγροτική πολιτική και πραγματικά θα είναι αυτά τα οποία θα είναι χρήσιμα και θα εφαρμόζουν το πρότυπο εφαρμογής που θα ακολουθήσουμε. Και τέλος, για τη νέα περιβαλλοντική δομή. Άκουσα κάποιες επικρίσεις σε σχέση με το πρασίνισμα. Έγινε κάποια παραπομπή σε αυτά που είπε το ελεκτικό συνέδριο. Νομίζω ότι η ανακοίνωσή μα ήδη κατά κάποιο τρόπο ανταποκρίνεται σε αυτό που είπε για το πρασίνισμα το ελεκτικό συνέδριο. Δηλαδή πρέπει να θεωρήσουμε το σύστημα. Θα πρέπει να έχουμε τρει διαφορετικέ έτσι, από τρει επιστρώσει, δύο ενδεχομένω, τρία επίπεδα, δύο που θα φορούν όλου του γεωργού στην Ευρώπη και μετά θα πρέπει να υπάρχει και ένα ευέλικτο εθελοντικό σύστημα σύστημα το οποίο θα αφορά και τον πρώτο αλλά και τον δεύτερο πυλώνα και το οποίο θα δίνει τη, στις χώρες την απαραίτητη ευελιξία ώστε να σχεδιάζουν περιβαλλοντικά μέτρα τα οποία θα ανταποκρίνονται στις τοπικές τους ανάγκες. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να βελτιώσουμε όλη την δομή της γεωργίας και της κοινή πολιτικής που όπως είδατε ότι στην, όπως λέμε στην ανακοίνωση, το μια από τις μεγάλες μας προτεραιότητες. Κατέγραψα επίσης και αυτά που είπατε πολλοί από εσά για, για, τα θέματα του, για τα θέματα του προπολογισμού και την κατανομή των κονδυλίων. Ξέρετε ότι εδώ έχουμε τις ε, προτάσεις του ΠΙΔΑΛΤΑΠΗ, προτάσεις που έχει ε, προγραμματίσει να καταθέσει η Κομισιόν στις 2 του Μάη, οπότε χρειαζόμαστε, χρειαζόμαστε για αυτό το θέμα, για τα δημοσιονομικά, δηλαδή λίγο χρόνο παραπάνω για να συζητήσουμε. Και τέλος για το θέμα του χρονοδιαγράμματος, του χρονισμού. Όπως είπαν προηγουμένως, η, η Κομισιόν προτίθεται να καταθέσει δημοθετικές προτάσεις τέλη του Μάη και από ό,τι είδα και εσείς θα ψηφίσετε την έκθεση στις 17 του Μάη. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή η σύμπτωση, κέρια, υποτενία δηλαδή ότι θα μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας όλες τις απόψεις όταν θα ολοκληρώσουμε ακριβώ τι νομοθετικέ μας προτάσει στην Κομισιόν και θα γνωρίζουμε ήδη από τις συζητήσεις που είχαμε τι γίνεται. Θα έχουμε δύο εβδομάδε ε, συζητήσεων και βεβαίω έχουμε κάθε πρόθεση να λάβουμε υπόψη μας τα, τις παρατηρήσεις και τι προτάσει. σα. Και τέλο να πω ότι κατέγραψα αυτό που αναφέρατε διάφοροι από εσά ω ανησυχία για την ανάγκη ύπαρξη μια μεταβατική περίοδου. Ξέρουμε ότι αφού οι συνομοθέτες υιοθετήσουν τους κοινού κανόνες για την γεωργική πολιτική, τότε ίσως να χρειαστούμε λίγο χρόνο ακόμα για να τα εφαρμόσουμε αυτά, επειδή το νέο πρότυπο εφαρμογής είναι πραγματικά νέο και θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στι χωρε μέλη για αυτό το νέο σύστημα, ώστε να είμαστε επιτυχεί. Θα διασφαλίσουμε λοιπόν ότι οι χώρες μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους αυτή την απαραίτητη χρονική περίοδο και ότι θα έχουν επαρκές περιθώριο να δουν ακριβώς ποιοι θα είναι οι νέοι βασικοί κανόνες και τι προσαρμογές πρέπει να κάνουν στα συστήματά τους. Νομίζω ότι βεβαίως θα διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρχει βιασύνη εδώ και ότι θα έχουμε ένα μοντέλο το οποίο πραγματικά θα είναι αποτελεσματικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θέλω καταρχά να ευχαριστώ του συναδέλφου. Θεωρώ ότι ήταν επικοδομητική η συζήτηση σήμερα. Πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα ακούστηκαν, οι προτάσει των συναδέλφων. Του ευχαριστώ θερμά. Βεβαίω δεν είναι δυνατόν τώρα να αναλύσω διεξοδικά τις 30 παρεμβάσεις, είναι και αργά. Θα πρέπει να είμαι σύντομος λοιπόν. Από αυτά που ακούω πάντως για το νέο μοντέλο, νέα σχέση, ε, ακούω να λέτε ότι δεν πρέπει να την προδικάσουμε εκ των προτέρων. Μπορούμε να δούμε τι μπορεί να προσφέρει η κοινή γεωργική πολιτική ε, με όσο το δυνατόν απλούστευση, αν μας το επιτρέπει αυτή η νέα σχέση, απλούστευση της γραφειοκρατίας αν μας το επιτρέπει όμως, γιατί κάποιες ε, από τις παρεμβάσεις που ακούστηκαν ε, έλεγαν ότι πρέπει με πολύ μεγάλη προσοχή να εξετάσουμε αυτή τη νέα σχέση και για την απλούστευση αλλά και για την γραφειοκρατία και για την ε, μετακύληση της πολιτικής, την επανεθνικοποίηση που ανέφεραν και πολλοί συνάδελφοι, αλλά και τις περιφερειακές αρμοδιότητες που θα πρέπει να εξετάσουμε. Βεβαίως, δεν ε, ισχυρίστηκα ότι η έκθεσή μου ήταν πλήρης, πλήρης ή ότι δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα. Πολλά είναι τα θέματα. Η δασοπονία, η, δασοπονια η ε, τα, οι απομακρυσμένες περιοχές, το Ποσέιντον που ακούστηκε, η μελισσοκομεία. Ήδη μόλις πρόσφατα καλύψαμε μια έκθεση, σε μια έκθεση το τομέα αυτών. Λοιπόν, δεν ήταν δυνατόν να καλύψω κάθε τομέα στην έκθεση αλλά ασφαλώς θα κατατεθούν τροπολογίες και πολύ ευχαριστώ θα τις συμπεριλάβω σε συνεννόηση πάντα με τους ε, συντάκτες τους στο κείμενο. Ε, βεβαίως, ακούω από τα όσα είπαν οι ότι πρέπει να είμαστε πιο ξεκάθαροι στο τι ζητούμε στην αρχιτεκτονική για το πρασίνισμα και πιο απαιτητικοί επίσης. Για τον κύριο Γιάρ, Μπορεί κανείς να διαβάσει τα πράγματα όπως τον βολεύουν, αλλά δεν είπα ότι η, αναλογικό, η αναλογική μείωση των ενισχύσεων και το ανώτατο όριο περνάνε στην εθνική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Δεν είπα εγώ κάτι τέτοιο. Είπα ότι θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η αναλογική μείωση παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο για το κάπινγκ είπα ότι πρέπει να περάσει στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Το ανέφεραν και άλλοι άλλωστε. Με αυτά θεωρώ ότι πολύ σωστά αναφέρθηκαν οι συνάδελφοι ε, στα σχόλιά τους, στην εθνική τους προοπτική, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και θα ακουστεί στη συζήτηση. Και επίσης για την κυρία Μαγκίνες θα επικαλεστώ τα λόγια της για να ολοκληρώσω ότι δεν πρέπει να εξολοθρεύσουμε την έκθεση με υπερβολικά πολλές τροπολογίες. Δεν πρέπει να λησμονούμε ότι οι τροπολογίες υπερβολικές μπορεί να περιορίσουν ε, μάλλον δεν θέλω να, ζητήσω να περιοριστεί η δυνατότητα για τους συναδέλφους ε, οι αρμοδιότητες και εξουσίες για διατύπωση τροπολογιών αλλά μην χάσουμε τελικά την ουσία της έκθεσης, μην καταλήξουμε τελικά σε ένα κείμενο το οποίο δεν θα εκφράζει το Κοινοβούλιο και την ε, πλειοψηφία των βουλευτών. Ε, παραλαμβάνω λοιπόν ότι πρόκειται για μια έκθεση η οποία πάνω απ' όλα ευθύνει ένα μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτάσεις και ιδέες, ενάβσματα που περιμένουμε ότι θα λάβει υπόψη. Εάν δεν το πράξει, τότε έχουμε δικαίωμα, πρωτοβουλία, έχουμε δικαίωμα νομοθετικό και βέβαια είναι μια αρχή αυτή την οποία δεν πρόκειται να λησμονήσουμε. Το απαραίτητο είναι να έχουμε μια σαφή θέση. Μια σαφή θέση έστω και αν δεν είναι υπερβολικά διεξοδική η έκθεση. Δηλαδή καλό είναι να μην χαθούμε στις λεπτομέρειες. Χρονοδιάγραμμα. Θα είναι δύσκολο, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, το αντιλαμβανόμαστε, ίσως και αδύνατον να ολοκληρωθεί στην τρέχουσα θητεία η μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής. Αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει ο στόχος μας να είναι να δουλέψουμε πάνω σε νομοθετικές προτάσεις και να τις ψηφίσουμε τις νομοθετικές αυτές προτάσεις. Εάν δεν επιδιώξουμε αυτόν τον ε, στόχο, τότε θα μπορούσαμε και να μην κουραστούμε με παραπάνω δουλειά. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να κάνει το κοινοβούλιο, να διατυπώσει το κοινοβούλιο μια θέση ε, στο τέλος της θητεία του, αν δεν την υποστηρίξει και με μια νομοθετική πρόταση. Α τα αφήσουμε για το επόμενο. Ιδάλω, μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά στο δεύτερο ήμιση του 18. Στόχος μου ήταν όχι να κάνω τη δουλειά μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα για την έκθεση αυτή για να την καταθέσω απλώς και μόνο. Ε, εγώ περίμενα ότι θα υλοποιηθεί και η προφορική τουλάχιστον δέσμευση του Επιτρόπου ε, που έλεγε ότι ψηφίζει το Κοινοβούλιο πρώτα και μετά καταθέτει νομοθετικές προτάσεις η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ψήφιση βέβαια του Κοινοβουλίου για μένα σημαίνει ψήφιση όχι στην Επιτροπή αλλά στην Ολομέλεια που είναι και η οριστική ε, διαμόρφωση του κειμένου. Αυτά. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, χρειάζομαι δυόμιση λεπτά για τον εαυτό μου να ευελιξία. Όχι Έχουμε το νέο μοντέλο λειτουργία, το New Delivery Model, το οποίο απαιτεί εργαλεία. Φυσικά όλα πρέπει να βρίσκονται υπό τον έλεγχο τη Επιτροπή. Ούτω ώστε να τηρήσουμε την αρχή μα περί ανταγωνιστικότητα. Φυσικά έχουμε και όλους τους αγαπημένους μας τομείς, τα μικρά αγροκτήματα και τα λοιπά τα λοιπά θα πρέπει να καλύπτει το 30% των αγροκτημάτων υπό τον πρώτο πυλώνα, ενώ το 70% πρέπει να σχετίζεται με τα θέματα μεικτής συμμόρφωσης, πολλαπλής συμμόρφωσης. Αν τηρήσουμε λοιπόν αυτό το 30% στο νέο μοντέλο και διατηρήσουμε και το 70%, τότε η πολλαπλή συμμόρφωση θα τηρηθεί. Και είμαι βέβαιος ότι αυτό θα γίνει κατανοητό και στα κράτη-μέλη. Καινοτομία, ναι, φυσικά είναι κάτι καλό για την ε, βιώσιμη γεωργία. Αλλά θέλουμε καλή καινοτομία, ψηφιοποίηση, άλλες ε, λύσεις, ε, λύσεις που ανήκουν σε μια νέα εποχή για τη γεωργία. Κάτι που θα βοηθήσει την ανάπτυξη των ε, αγροκτημάτων μας. Θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε νόσους, να αξιολογούμε την κατάσταση των φυτών κτλ. Να αντιμετωπίσουμε όλες τις νέες προκλήσεις και το θέμα της ε, ανανέωσης των γενεών ε, και της ε, στήριξης του εισοδήματος για τους γεωργούς και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε η κοινή γεωργική πολιτική δεν είναι μόνο για τους αγρότες, είναι για τους καταναλωτές, για το περιβάλλον. Όλοι τη χρησιμοποιούμε. Ε, μας προσφέρει και χαμηλότερες τιμές. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα θα εξαρτηθεί από την πολιτική βούληση, προφανώς. Εσείς ε, συμβάλλατε σε πολύ μεγάλο βαθμό, κάνατε πολύ σκληρή δουλειά. Έχουμε τον κανονισμό Omnibus που αποτελεί μια πολύ καλή λύση. Ανοίγει το ολοπεδίο, δημιουργεί δυνατότητες για νέες αλλαγές, τις διευκολύνει. Δεν χρειάζεται να επινοήσουμε από το μηδέν ε, μια νέα ε, κοινή πολιτική, απλά να τελειοποιήσουμε κάποια υπάρχοντα συστήματα. Θα ήθελα λοιπόν να απευθύνω έκκληση προς όλους τους συναδέλφους να υποβάλουν όσο το δυνατόν λιγότερες τροπολογίε. και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούει αυτή τη στιγμή τη συζήτησή μα, δεν χρειαζόμαστε λύσεις έτοιμε. ξέρουμε ποιοι είναι οι στόχοι. Υλοποιήστε του, εντάξτε του στι δικέ σα νομοθετικέ προτάσει στην Κομισιόν, διότι ξέρετε και του δικού μα στόχου. Το Νέο Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποκλείεται απλά να αναθεωρήσουν αυτή την ε, πολιτική, να την ε, αναδιατυπώσουν λίγο. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά τέλος πάντων, ε, τώρα μέχρι τις 19 Μαρτίου θα υποβληθούν τροπολογίες, στις 19 Μαρτίου θα οργανωθεί μια συνεδρίαση, οπότε ε, τελειοποιήστε τις τροπολογίες σας ε, μέχρι εκείνη την ημερομηνία ώστε να τις δώσουμε στην καλύτερη δυνατή τους μορφή και η συνεδρία της Επιτροπής θα λάβει χώρα στις 20. Ευχαριστώ πολύ. Μας έχει μείνει λίγος χρόνος ακόμα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και όλους εσάς. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό σας βράδυ και να ξαναευχαριστήσουμε φυσικά τον εισηγητή και όλους τους συνεισηγητές και τους συμμετέχοντες. Ευχαριστώ.